Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Κυρίως την κυρία Βλαδίσα Βλαντουλέσκου, η οποία είναι υπεύθυνη εργασίας ε, για το, της για τον έλεγχο ε, των όπλων και την εξαγωγή όπλων. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή συζήτηση λοιπόν με την ε, ε, έκθεση η οποία βασίζεται στο άρθρο 118 στα πλαίσια της προετοιμασίας της διαδικασίας εξέτασης του 2000, ε, του 2020 για το NPT και τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Σβέν ξένο εισηγητής, τον οποίων θα δώσω μετά το λόγο. Ε, εδώ αναφέρεται η θέση του Κοινοβουλίου ε, όσον αφορά την, δεύτερη, την δέκατη συγγνώμη, ε, εξέταση της διαδικασίας για τα πυρηνικά όπλα και της συνεδρίας που θα λάβει η χώρα την 19η Απριλίου του 2020. Η ε, η συνθήκη FNI έχει καταρρεύσει. Ε, επίσης απειλούνται άλλες ε, διαδικασίες και επομένως είναι θεμελιώδου σημασία σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να ξανασυζητήσουμε το NPT ε, έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί κοινό τόπο συζήτηση για τις διαπραγματεύσει και να γίνει ε, μία δήλωση ε, ουσίας η οποία θα μας οδηγήσει σε νέες διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τα τρία στοιχεία της συνθήκης. Επομένως, θα έχουμε πρώτα μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην πρότασή σα. και μετά η κυρία Βλαντουλέσκο θα μας ενημερώσει για τις προπαρασκευαστικές ε, εργασίες ε, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της προετοιμασία ε, για την διαδικασία NPT 2020 και επίσης για τα όσα θα ακολουθήσουν στο Consortium της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μη διάδοση των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 Ε, και θα συμμετάσχει στην συζήτησή μας. Επίσης, ε, να σας θυμίσω ότι η κυρία Μητσομίνα Καμίτσου ε, από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς επίσης και άλλοι εκπρόσωποι για τα πυρηνικά, επεδέχθησαν την πρόσκλησή μας για να συμμετάσχουν στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας και θα μας παράσχουν επιπλέον πληροφορίες για το NPT και συναφή θέματα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι συζητήσεις και οπωσδήποτε θα αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για επιπλέον στοιχεία ε, για την σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχει αλλάξει κάτι νομίζω όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση αυτή, για τη σύσταση αυτή. Ναι, μετά από την πρώτη εξέταση που θα κάνουμε σήμερα, ε, στις 28 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι, ε, θα ε, είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και στο Στρασβούργο 13 Φεβρουαρίου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών ενώ 19 και 20 Φεβρουαρίου θα έχουμε άφετ ε, και στην Ολομέλεια θα φτάσει στη δεύτερη του Ολομέλεια του Μαρτίου. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή έτσι ώστε να παρουσιάσει το σχέδιο σύσταση. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε αυτό το σχέδιο σχετικά με τη σύσταση ε, για την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της συνθήκης περί μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, την NPT. Είναι μια ε, πολύ σημαντική συνθήκη με στόχο την, ε, τον, τον να εμποδίσει την διάδοση των πυρηνικών όπλων και της πυρηνικής τεχνολογίας και να διαδώσει τις ειρηνικές χρήσεις της ε, Πυρηνική ενέργεια και να συνεισφέρει στον αφοπλισμό. Τρει στόχοι, λοιπόν, μη διάδοση, αφοπλισμός και ειρηνική χρήση. Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ τη δεκαετία του 70, το 1970 συγκεκριμένα, και φέτος εορτάζουμε την 50η επέτειο από τη θέση σε ισχύ η αρχική της ε, διάρκεια ήταν 25 χρόνια και μετά τα 25 χρόνια θα έπρεπε να γίνονται διασκέψεις επανεξέτασης κάθε 5 χρόνια. Ε, το μοντέλο που ακολουθήθηκε ήταν ότι δεν προέκυπταν αποτελέσματα σε κάθε, συνα... σε κάθε διάσκεψη, μάλλον σε κάθε δεύτερη διάσκεψη είχαμε κάποια αποτελέσματα. Το 2000 η διάσκεψη αναθεώρησης κατέληξε σε κάποιο αποτέλεσμα. Το 2005 δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Το 2010 κατέληξε στο σχέδιο δράσης των 64 σημείων και για τους τρεις πυλώνες της συνθήκης μετά το 2015 δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το σχέδιο κειμένου. θέτος η διάσκεψη αναθεώρησης θα γίνει τον Απρίλιο Και πέρυσι τον Απρίλιο έγινε μια συνάντηση προετοιμασίας ε, υπό την Προεδρία του πρέσβη της ε, Μαλαισίας στα Ηνωμένα Έθνη. 27 Απριλίου μέχρι 22 Μαΐου θα γίνει φέτος η διάσκεψη αναθεώρησης. Στην Υποεπιτροπή αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε κάποιες συστάσεις προς το Συμβούλιο και ολοκληρώσαμε τον Ιανουάριο το πρώτο σχέδιο έκθεσης, αρχές Ιανουαρίου δηλαδή. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε αυτό το σχέδιο σύστασης Στην υποεπιτροπή μα, 28 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για την τροπολογιών και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους σκιώδει εισηγητές το Φεβρουάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να εγκριθούν οι συστάσει στην Επιτροπή ΑΦΕΤ κατά τα τέλη Φεβρουαρίου και να συζητηθεί στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Πολύ σύντομα τώρα για το, περιεχόμενο των συστάσεών μας. Στο σχέδιο προτείνω να τονίσουμε τις βασικές αρχές ε, της πολυμέρειας ε, για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές ε, της διάδοσης πυρηνικών όπλων. Η συνθήκη NPT ήταν πολύ επιτυχημένη όσον αφορά τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων γιατί στα τέλη του 20ου αιώνα ε, υπήρχαν πολλές απειλητικές προβλέψεις με σενάρια αποκάλυψης, τα οποία δεν υλοποιήθηκαν σε σχέση με τη διάδοση των πυρηνικών όπλων. σύμφωνα με τη συνθήκη μπορούμε να αφαιρέσουμε τις ακραίες ε, υποθέσεις για να μπορέσουμε ε, να κάνουμε τις προβλέψεις μας και προβλέπω στην, ε, στο σχέδιο σύστασης να ενισχυθούν και οι τρεις πυλώνες της συνθήκης Ζητούμε από τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν τις βασικές αρχές για τη μη διάδοση και τον αφιπλισμό για να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα στο διεθνές περιβάλλον με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Ιδίως μιλάμε για μείωση του συνολικού αποθέματος πυρηνικών όπλων. Ζητούμε από τις Ηνωμένε Πολιτείε και τη Ρωσία που έχουν το μεγαλύτερο μέρος ε, του ε, πυρηνικού οπλοστασίου να αρχίσουν εκ νέου το διάλογο και ζητάμε από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να υποβάλουν μια δήλωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, και ε, στα όργανα που προβλέπονται από την NPT, στην οποία θα αναγνωρίζουν ε, τις υποχρεώσεις τους με βάση τη συνθήκη NPT. Εκφράζουμε τη λύπη μας για την κατάρρευση της συνθήκης INF. Και μιλάμε για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο τη ε, ε, της συνθήκης NPT σχετικά με την ε, αποστόχευση των πυρηνικών όπλων και την μη θέση τους σε συνεχή κατάσταση επιφυλακής. και τη μείωση των πυρηνικών όπλων όπως έχουν δεσμευθεί μετά το τέλος ε, του ψυχρού πολέμου. Κάποιοι είναι υπέρ μιας σταδιακής προσέγγισης και άλλα συμβαλόμενα μέρη πιστεύουν ότι θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά το πολιτικό κλίμα για να μπορέσουν να γίνουν οποιασδήποτε πρόοδοι προς την κατεύθυνση της βελτίωσης. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε να ωφεληθούμε από την ενίσχυση της συνθήκης NPT για να μειωθούν οι εντάσεις παγκοσμίω και να προχωρήσουμε προς τον τελικό μας στόχο ενός πλανήτη χωρίς όπλα. Προσβλέπω στη σημερινή συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες και με τους συναδέλφους και περιμένω τη δική σας συνεισφορά με πιθανές τροπολογίες στο σχέδιο συστάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Για να ξεκινήσουμε θα δώσω το λόγο στον Chris Πέκτερς για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω τη χαρά και τη τιμή σήμερα να αντικαθιστώ τον συνάδελφό μου, τον Αγνό Ντανζάν. Μόνο για σήμερα το πρωί θα συμβεί αυτό, αλλά για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να τον κάνω. Με έχει ενημερώσει και ο σκιώδης και έχω λάβει έξι σημεία, έξι σχόλια από τον συνάδελφό μου, τα οποία επιτρέψτε μου να διαβάσω. Επομένως, ο κύριος Ντανζόν ευχαριστεί, τον εισηγητή για την ποιότητα ε, της εργασίας του για αυτό το σχέδιο έκθεσης για ένα θέμα τόσο λεπτό, τόσο ευαίσθητο. Δεύτερον, θεωρεί ο κύριος Ντανζόν ότι το κείμενο αυτό σε αυτό το στάδιο είναι ισορροπημένο και αναπαριστά ορθά τα γεγονότα. Μας υπενθυμίζει τις αρετές της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων σε ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι όλο και περισσότερο τίθεται υπό αμφισβήτηση όλη η αρχιτεκτονική δομή της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του τρόπου ελέγχου αυτών, καθώς και ε, του αφοπλισμού διότι διαπιστώνουμε σιγά σιγά μια επιστροφή ε, των πυρηνικών τα οποία ξανέρχονται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά τις ε, στρατιωτικές αμυντικές στρατηγικές. Σύμφωνα με τον κύριο Ντανζόν, η προσέγγιση της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων σίγουρα δεν είναι η τελειότερη. Αξίζει όμως να οριμάσει, να είναι ρεαλιστική. Μας επιτρέπει να προβλέψουμε μέτρα και διατάξεις για την περιφερειακή και διεθνή ε, σταθερότητα και ασφάλεια. Είναι οικουμενική αυτή η συνθήκη και γίνεται αντικείμενο σεβασμού και τήρηση σε πολύ μεγάλο βαθμό, παρά τα όποια ασφάλματά της ή ε, ελαττώματά της. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα επιβιώσει στο δίνεκες και ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να τηρούν αυστηρά τις διατάξεις και τις ρήτρες της συνθήκης αυτής. Ο συνάδελφος, ο κύριος Ντόνζο, θα ήθελε να σας εφιστήσει την προσοχή στις ε, ανησυχίες που υπάρχουν σε σχέση με τη βούληση και τις πράξεις ε, το, της Ιρανικής πλευράς. Ξεκινά μια περίοδος αρκετής, ε, αρκετά μεγάλης αβεβαιότητας. Κατά πέμπτο λόγο χρειάζεται μια, ένας διεθνής στρατηγικός συντονισμός Φαίνεται ότι ξαναέρχονται τα πυρηνικά στο προσκήνιο και άρα η διεθνής αμοιβαία συνεννόηση υπονομεύεται σιγά σιγά. Είναι αναγκαίο και απαραίτητο να διατηρήσουμε όλες τις ρήτρε και τις διατάξεις τις υφιστάμενες για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και να έχουμε μια πολυμερή παγκόσμια τάξη η οποία θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Και τέλος, ο κύριος Ντονζό θα υποβάλει ε, τροπολογίες που θα κινούνται προς την κατεύθυνση των έξι αυτών βασικών παρατηρήσεων και σχολείων. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστούμε. Για το ΡΙΝΙΟΥ, ο μιλητής έχει φύγει, είναι εκτός αθούσης. Για τους πρασίνους λοιπόν δίνω το λόγο στον κύριο Σατορέ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ποιότητα της έκθεσης αυτής, η οποία είναι πολύ σημαντική, είναι ζωτική σημασία γιατί το θέμα είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια όλων μας. Επομένως κάνετε μια ποιοτική δουλειά και σας συγχαίρω για αυτή. Θα ήθελα να κάνω κάποιες συμπληρωματικέ παρατηρήσεις και να σας προειδοποιήσω για δύο πολύ συγκεκριμένου κινδύνους. Όντω επιστρέφουν τα πυρηνικά, αυτό υπόθηκε ήδη και η επιστροφή του ε, διαφαίνεται με αρκετά έντονο τρόπο. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, όλο και περισσότερες του κατά πόσο θα μπορέσουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις του, να προσφύγουν χώρες ε, στην ε, υιοθέτηση πυρηνικών. Αυτή η συνθήκη υιοθετήθηκε σε ένα πλαίσιο χρονικό κατά το οποίο ο κίνδυνος ήταν μεγάλος και προβλέπονταν και μέτρα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού σε περίπτωση έκρηξης για παράδειγμα. Δεν το λέμε τώρα για να αγχώσουμε τον κόσμο, όμως σε αυτό το νέο πλαίσιο από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι και να λαμβάνονται μέτρια αν ομιγέννητο συμβεί το δυστυχές να είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε στο μέγιστο βαθμό τον τοπικό πληθυσμό. Δεύτερο, που θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων. Ξέρετε, οι κυβερνοεπιθέσεις όχι μόνο από τρομοκρατικές ομάδες, ε, ε, ε, αποτελούν κίνδυνο. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος αυτός, υφιστάμενος. Και άρα πρέπει να έχουμε προβλέψει όλα τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας για να προλάβουμε την πυροδότηση πυρηνικών όπλων η οποία θα αποτελούσε αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης. Είναι ένας καινούριο κίνδυνος αυτός ο οποίος δεν υπήρχε όταν υπογράφτηκε αυτή η συνθήκη και θα πρέπει να λάβουμε αντίστοιχα μέτρα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη νέα συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τη στηρίζουμε όλοι δηλαδή αυτή, η οποία θα στηρίξει τον πυλώνα για τον αφοπλισμό της παλαιάς συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Αυτά λοιπόν είναι ε, τα θέματα που μας απασχολούν εμάς τους πρασίνους και θα υποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε επικοδομητικά σε ένα κλίμα που θα επικρατεί ο διάλογος και η πραγματική βούληση να έχουμε θετική ανταλλαγή απόψεων και ουσιαστική συμβολή για τη βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, για την ΑΕΔ, τον Πομφρίσκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συνθήκη με διάδοσης ε, πυρηνικών πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται ε, και κατά την άποψή μας να αποτελεί μάλιστα κεντρικό σημείο ρύθμισης ε, των πυρηνικών. Και εξ του συνάδελφου Ριβιέρ προτείνω στην Επιτροπή και στον εισηγητή, ε, ευχαριστώντας τον για την καλή εργασία, το εξή σημείο. Για περίπου μισό αιώνα η συνθήκη έδωσε τη δυνατότητα μη διάδοσης πυρηνικών και έδωσε τη δυνατότητα επίσης σε πολλές χώρες ε, να χρησιμοποιήσουν για ειρηνικούς σκοπούς ε, ε, τα πυρηνικά αλλά αυτή τη στιγμή διακυβεύεται ε, η ε, διεθνής ε, τάξη και λόγω της θέσης κάποιων χωρών, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Στην έκθεση ορθώς υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη στάση πολλών χωρών, οι οποίες τελικά αφαιρούν και αποδυναμώνουν τη συνθήκη και επομένως ενδεχομένως ε, την ε, διαδικασία αφοπλισμού. Οι χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουν την συνεργασία τους και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο. Και σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδυναμώσει τον ρόλο της. Βεβαίως κάθε χώρα έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τα ζωτικά της συμφέροντα και επομένως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με, τις, ε, ε, με τα όσα αναφέρονται στη σύσταση για πλήρη αποπυρηνικοποίηση. Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κίνα, ε, η Ρωσία είναι χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν τα πυρηνικά. Θα πρέπει να μελετηθεί πολύ προσεκτικά και η Συμφωνία της Γενέβης και η θέση του Ιράν. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2000 2011 ε, θα έπρεπε ήδη να είχε δημιουργηθεί μία μεγάλη ε, συμφωνία, συνθήκη κατά κάποιο τρόπο, συνασπισμός ε, κατά του, των απειλών του Ισλαμισμού και υπέρ των Ιουδεχριστιανικών ιδεοδών ο τρόπος ε, ε, χρήσης ε, όλων αυτών των όπλων θα πρέπει οπωσδήποτε να εξαρτάται από τον τρόπο συνεργασίας των χωρών. Κατά την έννοια αυτή θα υποβάλω και τροπολογίες. Ευχαριστώ. Très bien, merci. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εκπρόσωπος του Ρινιού. Κύριε Πασέσκου, έχετε ζητήσει το λόγο. Θέλετε Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ε, θέλω να σας ρωτήσω. Θέλετε να μιλήσετε για, την, ε, για το σχέδιο έκθεσης ή να κάνετε μια γενική τοποθέτηση. Ναι, ναι, όχι. Αφορά την έκθεση. Αφορά την έκθεση. Ως ε, ε, συνήθι, συνήθως ε, έχουμε θετικές λύσεις όσον αφορά θέματα εγγύησης της ειρήνης. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η επόμενη συνεδρίαση του μηνός Απριλίου δεν μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα, θετική έκβαση. Πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι προετοιμασμένη και για τα αρνητικά ενδεχομένως αποτελέσματα, αλλά και ε, για να ε, υποβάλει την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν τα πράγματα οδηγηθούν σε αρνητική έκβαση. Ωραία, καλό είναι να μιλάμε για πυρηνικούς κινδύνους, αλλά αν δεν πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα σε περίπτωση που δεν έχουμε αποτελέσματα το μήνα Απρίλιο, δεν κάνουμε τίποτα. Ε, εντάξει, εγώ είμαι απεσιόδοξος, ε, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά βλέποντας ε, και η συμμαχία Κίνας-Ρωσίας, ε, έχουμε την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ε, γιατί η Κίνα δεν θέλει να συμπεριληφθεί σε μια συνθήκη που θα εξισορροπήσει την ε, ε, ανάπτυξη των δυνατοτήτων που ανέπτυξε εκείνα τα τελευταία δέκα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα και για ενδεχόμενη αποτυχία μάλιστα της, ε, ε, του Απριλίου, της ε, συνάντησης του Απριλίου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχω και το κουράγιο, το θάρρος για να εκφράσω πραγματικά και υψηλοφόνο σε αυτά που σκέφτομαι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα σε σχέση με τη διάσκεψη του Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Βλαντουλέσκου, πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας ε, για την ε, μη διάδοση και τον έλεγχο των εξοπλισμών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκλησή σας. Και επιτρέψατε μου να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ καλή ε, έκθεσή του. Έρχεται σε πολύ καλή στιγμή αυτή η συζήτηση. Όπως ήδη ελέγχθη, το 2020 είναι πολύ σημαντικό έτος ε, για ε, το σύστημα της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων 50 ε, χρόνια μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης και 25 χρόνια μετά την επάπειρον παράτασή του και σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τις πολυμερείς συζητήσεις. Όπως ήδη ελέγχθη, το είπε και ο κύριος Μίξερ, οι διασκέψεις αναθεώρησης κάθε πέντε χρόνια νοούνται ως ε, επανέλεγχος του συστήματος και είναι ευκαιρία για τα συμβαλόμενα μέρη να συζητήσουν ε, σε αυτές τις συναντήσεις που βρισκόμαστε και προς τα που κινούμεθα. Ε, κάποιες συναντήσεις δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε τελικά αποτελέσματα. Αυτό συνέβη με την ένατη διάσκεψη το 2015 και γι' αυτό η φετινή διάσκεψη αναθεώρησης δεν πρέπει να αποτύχει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να μην υποκύψουμε σε τάσεις απεσιοδοξίας, αλλά να βρούμε κάποια κοινά σημεία συνεννόησης μετά από τις τέσσερις εβδομάδες της ε, διάσκεψης αναθεώρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως πεπισμένη ότι αυτή η πολύ σημαντική συνθήκη έχει πολύ μεγάλη αξία και την τωρινή χρονική στιγμή. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τις πολύ σημαντικές επιτυχίες της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας. με πολύ σημαντικά ε, θετικά στοιχεία για τον αφοπλισμό, δημιουργώντας και ένα στεναρό πλαίσιο για τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας. Υπενθύμησε σήμερα η Πρόεδρος, αλλά και οι κυρίες και κυρίες Ευρωβουλευτές, ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον ε, κλιμακούμενης έντασης. Υπάρχει διεθνώς ε, μία αρνητική ε, διάθεση όσον αφορά την αρχιτεκτονική της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και για τον έλεγχο των όπλων πέραν των όπλων μαζικής ε, καταστροφής. Και γι' αυτό θα πρέπει πολύ συνεκτικά να δουλέψουμε από την αρχή αυτών των, αυτού του κύκλου αναθεώρησης το 2017 και το 2018 η Ολλανδία και η Πολωνία που είχαν την Προεδρία των Επιτροπών έλαβαν πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουν ότι η, ε, ότι η διάσκεψη αναθεώρησης φέτος θα καταλήξει σε θετικά συμπεράσματα και η αποτυχία της διάσκεψης του 2015 ε, θεωρήθηκε σημαντική αποτυχία. Και πρέπει να αναστρέψουμε αυτή την αρνητική τάση και να βρούμε τώρα ε, ένα θετικό τρόπο προόδου το 2020. Έγιναν αρκετά workshops για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινέ θέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε την πρωτοβουλία και τον Απρίλιο του 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση 615 που υποστηρίζει τις δραστηριότητες που θα μας οδηγήσουν στην ε, τωρινή διάσκεψη αναθεώρησης. Η απόφαση του Συμβουλίου θέλει να υποστηρίξει διάφορες δραστηριότητες επικοινωνίας για την, ε, για το τι θα κάνει η διάσκεψη. Ο πρόεδρος της διάσκεψης αναθεώρησης μαζί με τα μέλη του Προεδρείου οργανώνουν και διεξάγουν διάφορες δράσεις. Εφτά αρκετά μεγάλες διασκέψεις τρία θεματικά σεμινάρια για τους τρεις πυλώνες της συνθήκης και τέσσερα περιφερειακά σεμινάρια στην Αφρική, Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, Ασία, Ειρηνικό και Μέση Ανατολή. Τρία από αυτά τα επτά σεμινάρια έχουν ήδη λάβει χώρα με σημαντικά αποτελέσματα. Με καλό κλίμα και με δέσμευση από όλου του συμβαλωμένου ε, στι περιφέρειε που αναφέρθηκαν. Έχουμε και άλλα σεμινάρια που θα ακολουθήσουν πριν από την διάσκεψη αναθεώρηση και αν θέλετε λεπτομέρειες μπορώ να σας ε, τις δώσω. Μια άλλη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι κάναμε ένα διάβημα που δεν έχει προηγούμενο, όπως και η απόφαση του Συμβουλίου ένα διάβημα προς όλα τα συμβαλόμενα μέρη, 189 συμβαλόμενα μέρη, όπου διευκρινίζουμε τη θέση μας και υποστηρίζουμε αυτό το πολύ σημαντικό κείμενο και ζητούμε από όλους να συμμετάσχουν στη συνάντηση της Νέας Υόρκης προσπαθώντας να βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις από όλους μαζί. Δηλαδή να αποφύγουμε τη δημιουργία μικροομάδων και να αποφύγουμε το κάποιες προτάσεις να κινούνται ταχύτερα από άλλες προτάσεις, ούτως ώστε να έχουμε μια συνολική συμβιβαστική λύση για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή αναθεώρηση της συνθήκης. Ο τρίτος τομέας δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι το Συμβούλιο μέσα στο 2020 και σίγουρα πριν από τη διάσκεψη αναθεώρησης θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα είναι ένα πολύ συνεκτικό έγγραφο και για τους τρεις πυλώνες με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προόδου. Το έγγραφο αυτό θα είναι ένα έγγραφο που θα προτείνει λύσεις και πρωτοβουλίες για το μέλλον για να αποφύγουμε τα τωρινά διέξοδα και το δύσκολο κλίμα στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτά ήθελα να σας πω και αν έχετε ερωτήσεις θα είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Ότ Κουβερτούρ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Όπως είπατε και εσείς, Θα ήθελα να κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις για το Consortium και όταν των όπλων και τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών. Είμαι επικεφαλής του Ιδρύματος για τη στρατηγική έρευνα και είχα ε, την αρμοδιότητα να οργανώνω τα, τις αιτήσει συναντήσεις του Consortium αυτού, το οποίο σίγουρα θα έχετε ακούσει. Το, η επόμενη μας συνεδρίαση ελπίζουμε, δεν είναι ε, οριστικό ότι θα λάβει χώρα στα τέλη Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου. Είναι μοναδική η στις αρχες ιουλιου ειναι μοναδικη στιγμη για τις 11 ε, χώρες που συμμετέχουν για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων να ανταλλάξουν απόψεις και να ενισχύσουν και να σφυριλατήσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα για τη μη διάδοση και για τον αφοπλισμό. Ελπίζω ότι πολλοί από εσά θα παραστούν σε αυτή τη συνάντηση που οργανώνουμε είτε τελειωνίου Ιουνίου είτε αρχέ Ιουλίου. Χρειαζόμαστε την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να ε, ενισχύσουμε τι ανταλλαγέ και την επικοινωνία και για το Κοινοβούλιο να έχει ισχυρή παρουσία σήμερα και τα επόμενα χρόνια. Αυτά καταρχά ω εισαγωγική παρατήρηση. Τώρα, λίγε σκέψει για το ιστορικό υπόβαθρο και το γενικότερο πλαίσιο. Το καθεστώ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων παγκοσμίω υφίσταται πιέσεις εδώ και πολλά χρόνια και αυτό αναπαρίσταται σε όλα τα σχετικά έγγραφα και εκθέσει που συντάσσονται από την αρχή αυτού του κύκλου αναθεώρησης. Εκτός από τις αγγείλε, αν θέλετε, το γεγονός ότι το 2010 είχαμε τη διάσκεψη για την αναθεώρηση και που έθεσε κάποια εισαγωγικά, δηλαδή ήταν μια παρένθεση αυτό, Είχαμε στη συνέχεια την άνοδο στην ε, κυβέρνηση του Ομπάμα που είχε μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα για τον αφοπλισμό στη διάσκεψη του 5 και του 15 αλλά και στη φετινή του Μαΐου ακολούθησαν τη συνήθη άγουσα ενώ η εκείνη ήταν η εξαίρεση. Και θα πρέπει να σας υπενθυμίζω ότι ε, από το 1975 μόνο πέντε αναθεωρητικές διασκέψεις έχουν καταλήξει στην υιοθέτηση τελικού κειμένου με συνένεση, με ομοφωνία που να έχει ουσία και νόημα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Αυτή την έκβαση της κάθε αναθεωρητικής ε, διάσκεψης ε, ε, πρέπει να τη θεωρούμε επιτυχία. Είναι αναπάντητο το ερώτημα αυτό, διότι η συνένεση εξορισμού μας οδηγεί στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Η υιοθέτηση ενός τελικού εγγράφου. Συνενετικά είναι επιτυχία επειδή εγκρίθηκε από όλου. Όταν ε, υπάρχει συνένεση, έχουμε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Έχουν συμφωνήσει στα ελάχιστα και αυτό μαρτυρά την αδράνεια, αν όχι την ακινησία. Ενώ για να επιβιώσει η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και να ε, ε, ε νοηματοδοτηθεί από μόνη τη, πρέπει να είναι δυναμική, πρέπει να δημιουργεί συνθήκε ασφαλεία επιτόπου. Υπάρχει σύγκρουση και αμφιλεγόμενε απόψει δηλαδή μεταξύ των κρατών μελών. Άρα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον όρο επιτυχία στα ε, πολυμερή φόρουμ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τώρα ε, την επέτειο για τη θέση σε ισχύ της συνθήκης φέτος, το Μάιο του 2020 και είναι ευκαιρία να τονίσουμε ότι η συνένεση δεν είναι ο, ο κανόνας ή το σύνηθες για τους ερευνητές για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η συνθήκη. Γιατί υφίσταται πιέσει η αναθεωρητική διαδικασία τη συνθήκη για τη μη διάδοση. Γιατί υφίσταται πιέσει στο καθεστώ το υφιστάμενο και υπάρχουν έξι παράγοντε που το πιέζουν. Πρώτον, έχουμε νέα κράτη αναδυόμενα στο διεθνέ σκηνικό που έχουν φιλοδοξίε, που τρέφουν φιλοδοξίε να γίνουν πυρηνικέ δυνάμει. και θεωρούν ότι όποιος έχει πυρηνικά έχει και δύναμη σαν κράτος και καλώς το θεωρούν γιατί ισχύει αυτό και ε, θεωρούν ότι είναι η καλύτερη δυνατή εγγύηση για την ασφάλεια. Ίσως το Ιράν, ίσως η Συρία και ίσως και άλλες χώρες οι οποίες σιωπούν αυτή τη στιγμή πιστεύουν κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα δεύτερον έχουμε τον εξυγχρονισμό της αναβάθμισης των οπλοστασίων αν θέλετε όλων των χωρών που έχουν ήδη πυρηνικά αυτός ο εξυγχρονισμός είναι ένα φαινόμενο που διαπιστώνεται τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια αναλόγως με τη χώρα για την οποία γίνεται λόγος. Τρίτον, οι μεγάλες πυρηνικέ χώρες δεν είναι πολύ ενθουσιώδεις ως προς τη διαχείριση του θέματος της διεθνούς ασφάλειας μέσω της πολυμερούς ε, προσέγγισης. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις της δεκαετίας του 90, οι οποίες έχουν ανασταλεί και το λέω αυτό κατεφημισμό και δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την Cut-Off Treaty, για τη συνθήκη αυτή. Και μετά έχουμε τη σχέση μεταξύ της μη διάδοσης και του αφοπλισμού στο πλαίσιο της συνθήκης για τη μη διάδοση και στο πλαίσιο της αναθεωρητικής διαδικασίας. Αυτή η σχέση δεν έχει σφυριλτατηθεί αρκετά, δεν έχει ενδυναμωθεί. Έχουμε τα άρθρα 2, 3 και 2 και 3 της συνθήκης που επιβάλλουν κάποιες προϋποθέσεις και έχουμε και το άρθρο 6 για τον αφοπλισμό. Αυτή η σχέση δηλαδή μεταξύ των δύο έχει αποδυναμωθεί, έχει χάσει την κινητήριο ισχύ του και έτσι τα κράτη-μέλη δεν εμπλέκονται δυναμικά στη βελτίωση της εφαρμογής του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα διμερή στρατηγικό εμπορικό διάλογο Ρωσίας-ΗΠΑ, ο οποίος χωλαίνει από την προσάρτηση της Κρυμαίας. Έχουμε ηγέτες που συμπεριφέρονται με τρόπο ο οποίος φαίνεται πραγματικά ανεύθυνος ε, στα μάτια της κοινότητας των χωρών που έχουν πυρηνικά και που, ε, ή όλων των χωρών που έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη για τη μη διάδοση. Από εκεί και πέρα. Έχουμε τη συμβατική και στρατηγική ε, ισχύ της Κίνας η οποία όλο και εντείνεται, όλο και αυξάνεται και η Κίνα στη διπλωματική της γλώσσα ε, τίθεται υπέρ της συνθήκης για τη μία διάδοση ενώ στο επιτόπου τελικά ακολουθεί άλλη άγουσα στο εσωτερικό της και στην πράξη. Σε, αυτές, σε αυτό το περίπλοκο πλαίσιο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει σε μια, σε μια δύσκολη θέση από την αρχή της δεκαετίας. Όλοι όλα αυτά αποτελούν ένα μικρό κόσμο για τη διεθνή ασφάλεια. Έχουμε τα πυρηνικά κράτη, τα μη πυρηνικά κράτη, τις μεσές δυνάμεις, τους ριζοσπάστες που είναι, τους ριζοσπαστικούς που είναι υπέρ της απόκτησης πυρηνικών, άλλους που θέλουν να χτίσουν γέφυρες ε, συνεννόησης και κατανόησης και ούτω καθεξής. Επομένως, είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες και πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει περισσότερα μέσα σε αυτό το πλαίσιο για τις συνθήκες για τη μία διάδοση από ό,τι έχει κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της. Να είμαστε ρεαλιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με τη συνένεση, με την ομοφωνία και το να βρεθεί ομοφωνία μεταξύ 28 κρατών μελών είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι ήταν τότε όταν υιοθετήθηκε αυτή η στρατηγική πριν από πολλά χρόνια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά δεν ασκεί τόσο μεγάλο επιρροή ε, ώστε να μπορεί να τροποποιήσει την πολιτική ασφαλείας των μεγάλων χωρών όπως η Ρωσία. Έχουμε το πείραμα της κατάρρευσης του INF πέρσι. Και αυτό έδειξε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν ό,τι μπορούσαν να πείσουν τη Ρωσία να τηρήσει τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της βάση της Ονθήκης και να, να πείσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αποσυρθεί από το, τη συμφωνία για το INF με το Ιράν, αλλά αποτύχε, ε, ε, έχει αποτύχει ε, η ευρωπαϊκή διπλωματία γιατί αποσύρθηκαν οι ή άλλως. Άρα δεν έπεισε κανέναν. Και σε αυτό το λεπτό ιστορικό πλαίσιο πρέπει να προσδιορίσουμε το ρόλο της Ευρώπης ως ε, αυτού που χτίζει γέφυρες μεταξύ των ε, ε, αντιθέτων πλευρών. Να διαδοθεί αυτή η αντίληψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παγκόσμιο στρατηγικό παίκτη, αυτό θα ήταν τεράστιο λάθος. Είμαστε ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εταίρο ο οποίος μπορεί να σφυριλατήσει επικοδομητικές συμμαχίε. Πρέπει να, η Ευρώπη να είναι επικοδομητικά επιθετική στην, ε, στο διεθνές ε, σκηνικό. Έχουμε ε, το υφιστάμενο πλαίσιο όπου υπάρχει απογοήτευση ε, ως προς την πολυμερή προσέγγιση. Δεν τη θέλει κανείς πια σε σχέση με 20 χρόνια πριν και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι υιοθέτησαν και επινόησαν τον όρο αποτελεσματική πολυμερής προσέγγιση. Τι σημαίνει αυτό ναι σε πολυμερείς λύσεις παρόλο που δεν είναι της μόδας και δεν γοητεύουν κανένα πια υπό τον όρο ότι ε, θα έχουμε αίσθηση ασφαλείας και μέτρα για την ασφάλεια επιτόπου στην πρακτική εφαρμογή εφαρμογή όλων αυτών. Η συνθήκη υπονομεύεται γιατί ο αφοπλισμός έχει έρθει σε τέλμα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την ενίσχυση της συνθήκης και την ενίσχυση των συνθήκων για να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 10 της συνθήκης, η ρήτρα για την απόσυρση, κρίσιμη σημασίας, είναι ένα από τα αδύναμα σημεία, από το αδύναμος κρίκος της συνθήκης μας. Για να αφιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερους πόρους ώστε να έχουμε τα δύο βασικά εργαλεία για τον αφοπλισμό, το CVT και το ε, δεύτερο. Για το πεδίο εφαρμογής λοιπόν ποιο είναι. Ε, να έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, να αφιερώσουμε τους πόρους μας σε ορισμένες πτυχές της στρατηγικής, τις πιο σημαντικές μόνο. Είναι ανοιχτό το ερώτημα. Θα ήταν χρήσιμο για όλα τα κράτη να καταλάβουν πόσο πολύ στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη μη διάδοση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ας δώσουμε νούμερα, αριθμητικά στοιχεία, αποτελέσματα. Θα, θα αναπαριστούν τα αποτελέσματα των δράσεών μας από το 2015, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε πετύχει. Και να σας υπενθυμίσω ότι η συνθήκη δράζεται σε τρεις πυλώνες. Το γνωρίζουμε αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε ξανά και ξανά. Ο τρίτος πυλώνας, οι ειρηνικοί χρήστες, άρθρο 4, δίνει λαβή ευκαιρία για μια πολύ επικοδομητική πρόοδο. Και στην πρόσφατη αναθεωρητική διάσκεψη, η οποία ήταν αποτυχία, θεώρησαν οι περισσότεροι, αυτό δεν ισχύει για τον τρίτο πυλώνα. Πρέπει να έχουμε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο αρμόδιο πολιτικό όργανο για να προωθήσει τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας, ε, ασφάλεια. Όλα αυτά είναι βασικοί στόχοι της Σύνθηκης για τη μη διάδοση. Είτε μας αρέσουν τα πυρηνικά είτε όχι, αυτό υπάρχει στη Συνθήκη. Άρα, όταν η κρίση είναι στρατηγική, σε τέτοιου είδους, σε είδους ε, χρονική περίοδο, μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε ε, με βάση αυτή τη διάταξη, με βάση τους τεράστιους πόρους που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιβεβαιώσουμε τη θέση μας και τα διαπιστευτήριά μας. Ίσως θα χρειαζόταν περισσότερη δημόσια διπλωματία, διπλωματία σε, στο δημόσιο λόγο. Δεν επικοινωνούμε αρκετά, δεν έχουμε πρόσβαση στο ευρύ κοινό έτσι ώστε να προβάλλουμε τα μηνύματά μας και πάνω σε αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε πιο εντατικά. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στον κύριο Σατουίπα που έχει ζητήσει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο παρεμβαίνοντας. Ήθελα να ρωτήσω το εξή για τη διάσκεψη του Απριλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινή θέση, συμφωνημένη θέση υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή θα πάει ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχοντας μια κοινή θέση. Επίσης, εάν και εφόσον υπάρχει, μπορείτε να μας δώσετε κάποιε λεπτομέρειες όσον αφορά το περιεχόμενο αυτή τη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Όχι. Ε, παρακαλώ πολύ. Ναι. Κοιτάξτε, είναι δύσκολη η ερώτηση. Δεν μπορώ εύκολα να την απαντήσω. Η απάντηση θα μπορούσε να είναι θετική, ναι, ναι, ε, έχουμε ε, πίστη ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια λεπτομερή και σαφώς εκπεφασμένη κοινή θέση. Έχουμε συμφωνημένες ε, κοινέ θέσεις σε προηγούμενες περιπτώσεις. Έχουμε ας πούμε αποφάσεις όπως τις λέγαμε παλιότερα ή συμπεράσματα πλέον του Συμβουλίου από το 2015. Δηλαδή παραδοσιακά έχουμε κοινή θέση όταν πηγαίνουμε ε, στην ε, κάθε φορά στην αναθεωρητική ε, ρεύκον. Προετοιμαζόμαστε πάντως, έχουμε ξεκινήσει ήδη την προπαρασκευαστική εργασία στο Συμβούλιο και για τους τρεις πυλώνες όπως αναφέρθηκε και εδώ, δηλαδή αφοπλισμός, μη διάδοση πυρηνικών και ειρηνική χρήση. Έχουμε θέσεις. Βεβαίως η θέση μας όσον αφορά την ειρηνική χρήση η θέση θα είναι πολύ πιο ε, συγκεκριμένη. Έχει ήδη συμφωνηθεί κοινή θέση με αναφορά σε όσα κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γενική Διεύθυνση GRC, DEVCO, Ενέργειας έχουν κάνει ε, πολλές προσπάθειες και καταβάλει πολλές, πολλούς πόρους τα τελευταία 5 με 10 χρόνια κατά την έννοια αυτή, δηλαδή όσον αφορά την ειρηνική χρήση ε, των ε, πυρηνικών. Βεβαίως, εμείς θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όρους που δεν είναι πάντοτε πολύ ε, δημοφιλείς αλλά έχουμε ε, εμπειρογνώμονες ε, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα θέματα ειρηνικής και μη ειρηνικής ε, χρήσης και επομένως στην αρχή της διάσκεψης εμείς ακριβώς θα επιστήσουμε την προσοχή σε αυτά τα θέματα. Έχουμε σίγουρα φιλόδοξο πρόγραμμα, δηλαδή θέλουμε να υποβάλουμε πλήρες πρόγραμμα για τον ε, αφοπλισμό, θέλουμε να ενισχύσουμε ε, την μη διάδοση και θέλουμε να προχωρήσουμε και όσον αφορά ε, τον πυλώνα του αφοπλισμού και ξέρουμε ότι υπάρχουν συμβαλόμενα μέρη της ε, συνθήκης μη διάδοση NPT που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο. Και εμείς θέλουμε να προτείνουμε πολύ απτά και συγκεκριμένα βήματα προς τη γραμμή αυτών που αναφέρατε προηγουμένως άλλωστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε... Ε, ναι, όχι, δεν νομίζω ήταν για μένα το, η ερώτηση, επομένως όχι, δεν θέλω να απαντήσω. Ο κύριος Μίξερ, παρακαλώ. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες για τα όσα μας είπαν. Αυτή η προσπάθεια συστάσεων είναι ε, πάρα πολύ σημαντική. Θα αποτελέσει άλλωστε και το input που θα έχουμε σε αυτήν την ε, ε, διάσκεψη. Βεβαίως, πιστεύουμε ότι ο έλεγχος των όπλων είναι ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει βεβαίως και την συνθήκη για τη μη διάδοση NPT και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το μελετήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ε, βέβαια είδαμε δυστυχώς ε, κάποιες άλλες ε, συνθήκες, ΑΕΝΕΦ και λοιπά να έχουν ε, αποτύχει. Απ' την άλλη μεριά έχουμε άλλες συνθήκες οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν, CTB και λοιπά. Έχουμε και την νέα συνθήκη για την κατάργηση των πυρηνικών που αφορά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ δεν το βλέπουν οι περισσότεροι πολύ ευνοϊκά. και άλλωστε και στην, στο προσχέδιο σύστασης αναφέρεται και ως μια γενικότερη επιθυμία της διεθνούς κοινότητας ε, για ελεύθερη, ε, ελεύθερο πλανήτη από τα πυρηνικά. member states. Uh, so there are Εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορές και μεταξύ μας και μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε μία εβδομάδα περίπου θα έχουμε και νέες συζητήσεις Αυτό που δεν θέλουμε σίγουρα είναι να εξισωθούν οι χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν σωστά τα πυρηνικά με χώρες οι οποίες ε, ε, έχουν προβληματική ε, χρήση. Επίσης μπορούν να υπάρξουν επικαλύψεις μεταξύ χωρών ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. και εν πάση περιπτώσει όσο υπάρχουν πυρηνικά στον πλανήτη ή ε, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ε, είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε ε, χρήση. Ναι, βεβαίως υπέρ της μη διάδοσης, ναι υπέρ της μείωσης και του πυρηνικού αφοπλισμού. Προς τα εκεί θα πρέπει να πηγαίνουν όλες οι προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες που μας διαφώτισαν σήμερα το πρωί και που μοιράστηκαν μαζί μας τόσα πράγματα, καθώς επίσης και για τον συνάδελφο. Λοιπόν, υπενθυμίζω, επόμενη Τρίτη, 28 ε, Ιανουαρίου, το μεσημέρι, ε, η εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Chers collègues, euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να ξαναρχίσουμε. Παρακαλώ, αν έχετε συζητήσεις, περάστε έξω για να μην έχουμε συζητήσεις μέσα στην αίθουσα. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε στην ώρα μας, όπως είναι και οι φιλοξενούμενες. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον στρατηγό Κλάουντιο Γκρατσιάνο, πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Στατιωτικής Επιτροπής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην Επιτροπή μας και περιμένουμε να ακούσουμε αυτό που έχετε να μας πείτε. Κατόπιν διαβούλευσης ε, με την εκπρόσωπο, το Κοινοβούλιο θέλει να ε, συζητά και να ενημερώνεται για τις διάφορες πρωτοβουλίες όσον αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες. Το σχέδιο πρωτοβουλίας ε, για την διαρθρωμένη συνεργασία διαμορφώνεται τώρα και στις συστάσεις θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει και τις συστάσεις των τελικών χρηστών για τη διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών. Η Συντηρητική Επιτροπή ε, εξασφαλίζει την συνοχή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίω η Υποεπιτροπή Ασφάλεια και Άμυνα, σα διαβεβαιώνει ότι έχετε την υποστήριξή μας και θα διαμορφώσουμε ε, ε, τις αντίστοιχες προτάσεις. Πάνω από 70% των Ευρωπαίων έχουν πει ότι τους ανησυχεί το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας και πρέπει να ανταποκριθούμε. Ε, στρατηγέ Γκρατσιάνο, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τα τελευταία συμπεράσματα ε, της Στρατιωτικής Επιτροπής στη σύνθεσή του με τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλή σας μέρα. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ στην Επιτροπή σας. Με τιμά η πρόσκλησή σας και θεωρώ ότι είναι και ένδειξη της σημασίας που αποδίδεται στην συνεισφορά της Στρατιωτικής Επιτροπής στην διάσταση της ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, η Στρατιωτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύω και την οποία εκπροσωπώ, Εκπροσωπείται 28 και σύντομα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέσω ε, ενό στρατιωτικού εκπροσώπου, του αρχηγού του επιτελείου ή στρατιωτικού εκπροσώπου η Στρατιωτική Επιτροπή προσπαθεί ε, να ακούγεται η φωνή του τελικού χρήστη των στρατιωτικών δυνατοτήτων, ώστε να ενημερώνονται ε, οι αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι απόψεις μας να ενσωματώνονται στις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ασχολούμαι με τη στρατιωτική δημοκρατία και είμαι και εκπρόσωπος ε, για θέματα ε, της Στρατιωτικής Επιτροπής προς τον, είπα, το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την αρμοδιότητα να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των ε, διαφόρων σεναρίων για τα οποία δίνουμε και την γνωμοδότησή μας. Για να μπορούμε να συζητήσουμε σωστά το θέμα των στρατιωτικών δυνατοτήτων, θα ήθελα να ξεκινήσω παρουσιάζοντάς σας την άποψή μου για την τωρινή κατάσταση ασφάλειας και άμυνας. Το νέο έτος δεν ξεκίνησε πολύ καλά, δυστυχώς. Οι επιθέσεις στο Ιράκ δεν ήρθαν ως έκπληξη. Γνωρίζαμε ότι υπήρχαν ήδη τα συμπτώματα εδώ και χρόνια. δεν ήρθαν σαν έκπληξη, αλλά πρέπει να δούμε τώρα ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα. Όλες αυτές οι κρίσεις μπορεί να έχουν πολλές επιπτώσεις και περιφερειακά, αλλά και για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Ένας επικίνδυνος συνδυασμός του φαινομένου της πεταλούδας με το φαινόμενο ντόμινο, όπου μια κρίση έχει συνέπειε σε άλλα μέρη του πλανήτη και μια κρίση δημιουργεί και νέες κρίσεις. Μιλάμε, μιλάμε για απειλές. Οι περισσότερες απειλές προέρχονται από τον Νότο, από τη Λιβύη μέχρι το Σαχέλ και μας υποχρεώνουν να εξετάσουμε ε, την ε, εξέτασή μας, ε, την στάση μας ε, για το τρίγωνο της αστάθειας. Ένα τρίγωνο που αποτελείται από την εξάπλωση της διεθνούς τρομοκρατίας σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων και των ε, ξένων μαχητών. Η μείωση της ασφάλειας λόγω της έλλειψης σωστής διακυβέρνησης. Υπενθυμίζω ότι το μέλλον της Ευρώπης αφορά και τη Λιβύη και χώρες, ε, γειτονικές χώρες όπως το Σαχέλ. Και ο κύριος Μπορέλ, είπα εκπρόσωπος, αποδίδει μεγάλη σημασία ε, στην ε, περιοχή αυτή. Προσπαθούμε να έχουμε ένα νέο ρόλο στην περιφέρεια αυτή εξετάζοντας και τη συμμετοχή των άλλων χωρών όπως η Ρωσία, Τουρκία ή και Κίνα που προσπαθούν να καλύψουν κενά που έχουν αφήσει κάποιοι άλλοι. Για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχει ανάγκη ταχείας αντίδρασης πριν φτάσει η κατάσταση σε ένα σημείο μη επιστροφής. Το ερώτημα είναι ποιος λαμβάνει την πρωτοβουλία. Είναι προφανές ότι κανένα κράτος μόνο του δεν είναι σε θέση και δεν νομιμοποιείται να αναλάβει όλες τις προκλήσεις χωρίς να έχει και κανένα δευτερεύοντα στόχο. Θα πρέπει λοιπόν οι ευθύνε να βαρύνουν τη διεθνή κοινότητα και μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτείται λοιπόν όχι μόνο μία προσέγγιση όπου θα αντιδρούμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά και θα είμαστε ενεργά συμμετέχοντες. Και γι' αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό ως Ευρωπαϊκή Ένωση. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμφανιστεί ως παγκόσμιος ε, παράγων, ως ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό πρέπει να δρούμε αποφασιστικά και για να αποφύγουμε κενά ασφάλειας. Να μην γίνονται στόχοι μεμονωμένων παραγόντων τα κενά που αφήνουμε εμείς. Αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιώντας πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά μέσα την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την ονομάζουμε, θα πρέπει να δράσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ως πάροχος ασφαλείας διεθνώς, δρώντας είτε αυτόνομα είτε ως εταίρος μέσα στο ειλικρινές πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας. Ιδίως όταν οι κρίσεις αυτές αφορούν τους ε, κοντινούς μας γείτονες. Βέβαια, μιλώντας ως στρατιωτικός, πιστεύω ότι οι κρίσεις αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα μόνο από αυτά τα μέσα που προανέφερα, αλλά με μια ισορροπημένη προσέγγιση. Η πρόσφατη ιστορία μας διδάσκει εξάλλου ότι όταν αναζητούμε διπλωματικές λύσεις, συχνά πρέπει να δημιουργούμε ένα πλαίσιο ασφαλείας χρησιμοποιώντας στρατιωτικά μέσα, τουλάχιστον ως ένα παράγοντα ε, ενίσχυσης για να μπορέσουμε να δράσουμε. Δεν υπάρχει μόνο η στρατιωτική λύση για την τωρινή κρίση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να βρεθεί λύση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτικά μέσα, τουλάχιστον για να μας διευκολύνουν. Μιλώντας για στρατιωτικά εργαλεία, αυτό δεν σημαίνει ε, ότι ε, θα εμπλακούμε σε μάχες, αλλά θέλουμε να, να δράσουμε συμπληρωματικά για να υποστηρίξουμε τις διάφορες ε, φάσεις της κρίσης, ώστε να αποκλιμακώνονται οι κρίσεις και να επανερχόμαστε στην πραγματικότητα. Ο ίδιος εκπρόσωπος είπε πριν από δύο μέρες ότι δεν μπορούμε απλώς να κηρύξουμε εκεχηρία και να φύγουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες προστασίας και παρακολούθησης. Και μάλιστα ενδεικτικά αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σκέφτεται κάτι το οποίο και εγώ υποστηρίζω, να επανενεργοποιήσει την επιχείρηση Σοφία με όλα τα πιθανά μέσα για να ενισχύσουμε ε, το εμπάργκο των ε, όπλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει ένα σαφές ε, μήνυμα συνοχής και αποφασιστικότητας αναγνωρίζοντας την ανάγκη του κατεπήγοντος που πολλές πλευρές αναφέρουν. Αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι τώρα, έτοιμοι να δράσουμε τώρα ή και στο μέλλον, είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε τις δυνατότητες ε, ε, των αποστολών. Θα πρέπει να δείξουμε ενότητα στην προσέγγισή μας σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, παραδείγματο χάρη, για τη βελτίωση με όλους τους παράγοντες που θέλουν να, να δράσουν με συνέργεια για να επιτύχουμε τους κοινούς στόχους. Αλλά για να είμαστε αξιόπιστοι πάροχη βοήθειας και για να μπορούμε να υποστηρίξουμε το δικό μας σενάριο αν απαιτείται, πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα και δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο για τις, με τις πρωτοβουλίες και τα μέσα ασφάλειας και άμυνας. Υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως η PESCO, η CARD, η DP και η EDF. Έχουμε εργαλεία τα οποία είναι μοναδικά για την παρακολούθηση των, και τον προγραμματισμό των αποστολών μας. Χρειάζεται βέβαια η δέσμευση των κρατών μελών για να τα επιτύχουμε όλα αυτά, για να έχουμε μια αξιόπιστη προσέγγιση. Το EDF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, ε, έχει ε, βρει μεγάλη ανταπόκριση. Έχουμε ένα μηχανισμό που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μέσα και οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο της έρευνας για να μπορούν να συμμετέχουν τα κράτη-μέλη εφόσον γίνεται η συμμετοχή τους περισσότερο ελκυστική. Θέλουμε να αποφύγουμε τη σπατάλη πόρων και την επικάλυψη προσπαθειών. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το EDF αποτελεί τη βάση για να κρατήσει η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία την τεχνογνωσία και τις ερευνητικές δυνατότητες που αποτελούν πρωτοχική σημασίας μέσα για την μακροπρόθεσμη επιβίωσή της. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα, το EDF, αποτελεί έναν παράγοντα που θα προωθήσει την καλύτερη συνειδησία, γιατί σε αυτό το τομέα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες δεν είχαν κάνει κάτι. Και πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία επιτυγχάνουμε με το EDF θα είναι χρήσιμα και για το ΝΑΤΟ, γιατί αυτά που είναι καλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σωστά και για το ΝΑΤΟ ως δυνατότητες. Είναι ένα ορόσημο λοιπόν το EDF για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία από τις καλύτερες επενδύσεις ε, για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε ούτε καν να, διανοηθούμε να περικόψουμε τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, ιδίως στην παρούσα ιστορική στιγμή. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ε, την αξία όλων αυτών των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας για να έχουμε αυτά αποτελέσματα από τα τωρινά μέσα πριν προωθήσουμε νέα μέσα. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω το σημαντικό ρόλο του στρατιωτικού τομέα. Καταρχήν σε στρατηγικό επίπεδο, διότι παρέχουμε τη συνεχή μας τεχνογνωσία και τις συμβουλές μας που είναι κέρια σημασίας για τη λήψη αποφάσεων από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Δεύτερον, ως κύριοι χρήστες, χρήστες των ε, ε, εργαλείων τα οποία παρέχονται από τις διαδικασίες αυτές. Αυτό βέβαια μας ε, αναθέτει μια επιπλέον ευθύνη. Αλλά τις ευθύνες αυτές τις αναλαμβάνουμε ευχαρίστως, ακριβώς λόγω της μεγάλης μας τεχνογνωσίας και γνώσεων του τομέα. η Στρατιωτική Επιτροπή ασχολείται με πρωτοβουλίες όπως η ΠΕΣΚΟ ή η ΚΑΡΔ. Όταν μιλάμε όμως για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, αυτό δεν ισχύει ακόμη. Μια αλλαγή για τη Στρατιωτική Επιτροπή θα ήταν να είναι περισσότερο παρούσα στο EDF υπό την, τον τωρινό σχηματισμό της για να παρέχει συμβουλές. Η Στρατιωτική Επιτροπή παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να συμβάλλει για να βοηθήσει τους λαμβάνοντες αποφάσεις. Έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Γνωρίζουμε τη σημασία που έχει η προσπάθειά μας για όλες τις στρατιωτικές δράσεις και συνεχίσουμε μέσω των δράσεών μας να προσφέρουμε στην μεγαλύτερη ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ συλλογικών προσπαθειών και ευθυνών του, κυρίαρχου, του κάθε κυρίαρχου κράτους για να μπορέσουμε να έχουμε το απαραίτητο επίπεδο στρατηγικής αυτονομίας και για να μπορούμε ταυτόχρονα να μιλάμε με μία και μόνη φωνή. Το να έχουμε δυνατότητες στη διάθεσή μας θα συνεισφέρει στο να ολοκληρώνουμε το στόχο μας καλύτερα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ρόλο όχι μόνο εκπαίδευσης αλλά και παρακολούθησης ε, και ένα συνοδευτικό ρόλο. Αυτό και για τις εκπαιδευτικές αποστολές μας αλλά και για την αποστολή στη Σομαλία. Αυτό βοηθάει βοηθά και τις δυνάμεις επιτόπου, αλλά και δίνεται η εικόνα της ε, πιο, πιο έντονης συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, διεθνή κοινότητα και έναντι των στρατηγικών μας ανταγωνιστών. Επιπλέον, οι αποστολές μας γίνονται πιο αποτελεσματικές και αυτό θα δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να συνεισφέρουν περισσότερο σε αυτές τις αποστολές και να καλύπτεται και το τωρινό έλλειμμα προσωπικού. Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και τους άλλους διεθνείς εταίρους βέβαια. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για τα θέματα αυτά. Ελπίζω να σας έδωσα μια εικόνα για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις τρέχουσες υποθέσεις. Θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι οι εμπειρογνώμονες σε στρατιωτικά θέματα πάντοτε είναι διαθέσιμοι για να παρέχουν συμβουλές και η εμπειρία μας είναι πάντοτε στις υπηρεσίες αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις. Η παρουσία μας τόπου είναι ανεκτήμητη σημασίας. Άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε και όλους τους αξιότιμους ε, βουλευτές και θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ στρατηγέ. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στο συντονιστή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τον κύριο Μίξεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, στρατηγέ, για την πολύ ολοκληρωμένη και περιστατωμένη σας παρουσίαση. Έχω κάποια ερωτήματα να σας απευθύνω, που προέκυψαν ε, από το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ψηφίσαμε την ετήσια έκθεση. Ένα από τα βασικά θέματα ήταν η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συζητούμε γενικά τι σημαίνει αυτός ο όρος και στην Επιτροπή μας αλλά και στην Ολομέλεια. Και η συζήτηση ήταν πολύ τεταμένη. Δεν υπάρχει μεγάλη συνένεση για το τι ακριβώς σημαίνει στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή και κατά πόσο υπάρχουν όρια σε αυτήν την επιδίωξη. Όλοι, κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει ο όρος στρατηγική αυτονομία να ατύχει περιοριστικού ορισμού και όχι ευρύ ορισμού. Με την έννοια ότι θεωρούν ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε απολύτως αυτόνομα έναντι του ΝΑΤΟ όταν ε, παρεμβαίνουμε στρατιωτικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω. Κατά δεύτερον, ως προς τις επιχειρήσεις, τις αποστολές τις οποίες επικουρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως προς αυτό. Έχουμε συμβάλει και έχουμε βοηθήσει στην επίλυση διαφόρων κρίσεων. Έχουμε τις ε, Εκπαιδευτικέ αποστολέ, συμβουλευτικέ αποστολέ, οι οποίες είναι τρέχουσες και διατηρούνται στο δινεκές ε, και στο Ιράκ και στην Αφρική. Αυτά τα συζητούσαμε εχθές και υπόθηκε ότι στο μέλλον όταν ε, εμπλακούμε σε επιχειρήσεις εκπαιδευτικές ή συμβουλευτικές, πρέπει να υιοθετούμε λύσεις ε, σύμφωνα με τις οποίες, που να είναι έτσι διαμορφωμένες δηλαδή, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει τους πόρους για την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική υπηρεσία, αλλά η δύναμη προστασίας επιτόπου να αποτελεί αντικείμενο συμμαχίας μεταξύ των στρατών ορισμένων χωρών μελών και όχι ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ως Συμμαχία Κρατών για την Προστασία και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβουλευτική και εκπαίδευση μόνο. Έτσι να μοιραστούν αυτά τα τρία σκέλη, γιατί θεωρούν ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό. Υπάρχει αυτή η πρόταση. Ποια είναι η άποψή σας ε, για, το, ε, για την Αφρικανική Ήπειρο και για αυτή την ε, κατεύθυνση, αλλά και για άλλες περιοχές. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε και άλλους βολευτές που θέλουν να σας δώσουν ερωτήσεις και μετά θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Για το έλκο ο Κρίς Πέτερς παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έπρεπε να πάω σε άλλη επιτροπή για να ψηφίσω και γι' αυτό καθυστέρησα και δεν ήμουν εδώ στην αρχή της ομιλίας σας. Πολύ χαίρομαι, διότι ο συνάδελφος ε, θέτει ε, αυτό το θέμα το οποίο συζητήσαμε για το τι εστίστε Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία και αναφέρθηκε και στην έκθεση που ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Αγαπητέ στρατηγέ, ελπίζω ότι έχετε διαβάσει αυτό το τμήμα της έκθεσης, την παραγράφο η οποία αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία. Ε, δίδει μια πολύ σημαντική απάντηση για το τι πιστεύουμε για αυτό το ζήτημα. Είναι από το σημείο 20 και κάτω. Θα ακούσω βέβαια την απάντησή σας στον συνάδελφό μου γιατί είναι πολύ σημαντική αλλά η άποψή μας απεικονίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σημείο 20 και κάτω της εκθεσής αυτής. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Αμυντικό, Αμυντικό Ταμείο είναι πολύ σημαντικό. Ερωτώ λοιπόν, ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτού του ταμείου και της... Ε, και αυτό που κάνετε εσείς στην ε, Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει άμεση σύνδεση. Δεν έχετε τη δυνατότητα να προτείνετε project και σχέδια άμεσα. Πρέπει να τα περάσετε μέσα από το Συμβούλιο. Δεν... Ε, μπορείτε κατευθείαν να συνδεθείτε με το Ευρωπαϊκό ε, Αμυντικό Ταμείο και να πάρετε χρηματοδότηση από εκεί. Όντω έτσι ισχύει και αν ναι, ποια είναι η θέση σα, ποια είναι η άποψή σα. Ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ, κύριο Μπασέσκο, παρακαλώ. ενα από του κινδυνου που αναφέρατε, ε, στρατηγέ, και συμφωνώ άλλωστε μαζί σα ε, είναι αυτό το θέμα των ρευμάτων μετανάστευσης δηλαδή μετανάστευση κατά ρεύματα. Είναι προφανές ότι εάν περιοριστούμε όπως το παρελθόν μονάχα σε παρέμβαση στην ε, ε, Μεσόγειο για να σώσουμε ζωές, ε, στην Μεσόγειο πάντα, οπωσδήποτε θα συνεχιστεί το φαινόμενο αυτό, γιατί δεν θα το έχουμε εκριζώσει και τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο περίπλοκα. Κατά την ε, δική μου άποψη, το ε, για να ελεγχθεί η παράτυπη μετανάστευση σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν τρία πράγματα σε επίπεδο και ε, ε καλής, για να μην πω εξαιρετική συνεργασίας πολιτικής ανάμεσα στην στρατηγική και μη ηγεσία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις κύριες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι παράτυποι μετανάστες. Δεύτερον, θα πρέπει να παρέμβει και η ε, ε, οι υπηρεσίες ε, κατασκοπίας και οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με τους διακινητές, να αποκαλυφθούν οι διακινητές, γιατί για να περάσει κανείς, για να περάσουν την, διασχίσουν την Μεσόγειο, αυτοί οι μετανάστες πληρώνουν πάρα πολύ ψηλά ποσά σε αυτούς τους διακινητές που καμιά φορά είναι και έμποροι ανθρώπων, ασχολούνται δηλαδή και με το τράπεζο ε, γιατί εάν δεν καταφέρουμε να εκριζώσουμε αυτές, αυτά τα δίκτυα των διακινητών, ε, ε, τα οποία δίκτυα γίνονται ανεκτά από τις χώρες στις οποίες τα δίκτυα αυτά κινούνται, δεν θα καταφέρουμε κάτι. Ε, εάν σταματήσουν, εάν διαλυθούν αυτά τα δίκτυα των διακινητών, ε, τότε υπάρχει μία ελπίδα να, σταματήσει, ε, να σταματήσουν αυτά τα ρεύματα της παράτηψης ε, μετανάστευσης. Επίσης, όσον αφορά την διάσωση των ανθρώπων, βεβαίως είναι διεθνής υποχρέωση να διασωθούν άνθρωποι των οποίων η ζωή κινδυνεύει. Ναι, λοιπόν, είναι ε, σημαντικό το θέμα λοιπόν των επαναπροωθήσεων της διάσωσης αλλά ε, και της ε, διάλυσης των διακινητών και οπωσδήποτε όλα θα πρέπει να ξεκινήσουν και από τις σχέσεις με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι παράτυποι μετανάστες. Πρέπει να σταματήσουν τώρα αυτές, αυτά τα ρεύματα γιατί διαφορετικά θα γίνει πραγματική απόβαση. Όλα τα... Ε, το, το αναφέρει άλλωστε και μία πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να αναπτύξουμε συστηματική διαδικασία η οποία θα ξεκινάει από τη διπλωματική συνεργασία ε, που θα επιτύχει δηλαδή συμφωνίες επαναπροώθησης ε, με τις ε, χώρες αυτές. Θα πρέπει δε, όπως είπα και προηγουμένως, να διαλύσουμε τα συστήματα των διακινητών σε συνεργασία και με τις χώρες εντός των οποίων λειτουργούν αυτά τα δίκτυα. Ευχαριστώ, κυρία Μπονφρίσκο. Καλημέρα, στρατηγέ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, καθώς επίσης και για το ευρύ πλαίσιο το οποίο ε, μας παρουσιάσατε. Ζητώ συγγνώμη, συνάδελφοι, και ζητώ συγγνώμη και από την Προεδρία, γιατί ενδεχομένως δεν θα, είμαι, δεν θα μπορέσω να παραμείνω για να ακούσω τις απαντήσεις σας, αλλά θα τι διαβάσω βεβαίως. Συμφωνώ μαζί σας ο ρόλος ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς ε, αυτό, το, να παίξει δηλαδή το χαρτί της στρατηγικής αυτονομίας και της περιοχής που παρέχει ασφάλεια και απέναντι στην κλιμάκωση που διαπιστώνουμε τον τελευταίο καιρό και στην μεγάλη γεωπολιτική αταξία, η δικιά μας διαδικασία επιτήρησης, ελέγχου, κατάρτισης, παροχής ε, βοήθειας ακόμα και στρατιωτικής μορφής, ε, πραγματικά η συμβολή μας, λέω, μπορεί να είναι ε, μεγάλη και να αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία. Εγώ συμφωνώ όμως και με τις παρατηρήσεις που μόλις ανέφερε ο συνάδελφος Παντέσκου ε, και στα όσα πολύ ορθά ανέφερε ο κύριος Μπαντέσκου, ε, προσθέτω ότι η Σοφία ε, έδειξε τα όρια της στην ουσία. Ήταν αποτυχημένη επιχείρηση, αλλά εάν ε, στο μέλλον ασχοληθεί περισσότερο με την ασφάλεια των συνόρων μας και την ασφάλεια ε, εις ε, το, στη Μεσόγειο που αποτελεί κλειδί για την προστασία των πολιτών της Ευρώπης, τότε θα γίνει ένα εργαλείο σημαντικό. Όμως, επί του προκειμένου, ο ρόλος της Επιτροπής μπορεί να γίνει πιο προφανής κατά την, άποψή μας ε, χρησιμοποιώντας το αμυντικό ταμείο γιατί διαφορετικά ε, θα είναι ένα εργαλείο το οποίο γεννιέται με πολύ κακούς ιονούς. Ε, και σε μια ιστορική στιγμή όπως αυτή την οποία διανύουμε είναι και αντιιστορικό και αντιοικονομικό ε, να προωθήσουμε μια τέτοια θέση για αυτήν την ε, Επιτροπή. Νομίζω ότι και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου θα έχουμε την δυνατότητα και θα, θα βρούμε τον τρόπο να λειτουργήσουμε σωστά και σε σχέση με το Ταμείο αυτό. Η αποτελεσματική λειτουργία κατά την άποψή μου μπορεί να ε, και πρέπει μάλλον ε, να υλοποιηθεί με την δική σας επίβλεψη, με δικό σας μεγάλο ρόλο, με δική σας διαβούλευση έτσι ώστε να μην υπάρξουν επικαλύψεις, να μην υπάρξουν ε, να μην υπάρξει διασπάθηση χρημάτων και επίσης να μην υπάρξει μία πολυμέρεια όσον αφορά την αντίδραση τη στιγμή που πρέπει να υπάρχει αντιθέτως επικέντρωση της αντίδρασης. Τι άλλο μπορεί να κάνει η Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγκουίλα, παρακαλώ. Αγγιλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση να απευθύνω στο στρατηγό. Καταρχάς, ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στρατηγέ για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Κατά τη γνώμη σας, θα ήθελα να γνωρίζω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, το εγγύς μέλλον, ως προς την άμεση συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ερώτησή μου και θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που έθιξαν το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στη Μεσόγειο με την παράνομη μετανάστευση. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που πλήττεται, που υφίσταται αυτό το φαινόμενο. Δεν είμαστε αρκετά πλούσια χώρα για να μπορέσουμε να θρέψουμε όλους τους παράνομους μετανάστες, λέει ο Μιλήτρη, που φτάνουν στην ε, ε, πόρτα μας. Μη ζουν στο δρόμο κάθε μέρα και υπάρχουν και σε αυτούς τους παράνομους μετανάστες οι οποίοι αν θέλετε θέλουν να βρουν μια καλύτερη ζωή, αλλά με αυτούς έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν το κακό και παρισφρίουν δηλαδή στις ομάδες των μεταναστών και κακοποιά στοιχεία τα οποία ε, έχουν άλλες επιδιώξεις και άλλες βλέψεις, δυστυχώς. Ε, θα πρέπει να είναι εξατλητικός ο έλεγχος, δεν είμαστε πλούσια χώρα, και δεν ταιριάζει η Αφρική στο δικό μας έστω, έθνος. Χρειαζόμαστε πιο εξαντλητικούς ελέγχους και σας ευχαριστώ πολύ ε, που με ακούσατε και σας ευχαριστώ για την ε, παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στρατηγέ, πριν σας δώσω το λόγο, θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Επιτρέψτε μου και εγώ να σχολιάσω με την ιδιότητά μου της Προέδρου. Είπατε ότι επιθυμείτε να θελήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευρύνει την εντολή της στο Σαχέλ, στη Σομαλία, μεταξύ άλλων, να μην έχουμε μόνο εκπαίδευση, αλλά πλαισίωση και συνοδεία των τοπικών δυνάμεων. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των κρατών μελών προς το παρόν, τις γνωρίζετε. Χθες το πρωί Είχατε μια μακροσκελή συνεδρίαση για το Σαχέλ, για αυτή την περιοχή και όλοι είχαμε εμείς ε, σήμερα, το, χθες το πρωί, όλοι ε, αποκόμισαν την αίσθηση ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα και γρηγορότερα. Σημερίζονται την άποψη αυτή τα κρατημέλη, γιατί αυτό προέκυψε από τη χθεσινή μας συνεδρίαση για το Σαχέλ. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για την Ειρήνη είναι ένα εργαλείο χρήσιμο. Ποια είναι η γνώμη σας. Αυτό το μέσο, το χρηματοδοτικό, ποια είναι η θέση των κρατών μελών. Είναι ένα έργο το οποίο προγραμματίζεται από το 2018 και καλό θα είναι να πραγματοποιηθεί σύντομα. Έχετε το λόγο στρατηγέ. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σημαντικές ερωτήσεις που χρειάζονται μεγάλη ανάπτυξη και για κάποια από αυτά τα ερωτήματα δεν έχω και αρμοδιότητα να απαντήσω ως προς την πολιτική τους διάσταση. Να ξεκινήσω με τη στρατηγική αυτονομία που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην παγκόσμια στρατηγική γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πυλώνας, αλλά η έννοια της είναι πολύ πιο απλή. Είναι ένας πυλώνας αξιοπιστίας. Δεν μπορεί να υπάρχει παγκόσμια στρατηγική, δεν μπορεί κανείς να γίνει παγκόσμιος πάροχος ασφαλείας χωρίς να έχει στρατηγική αυτονομία που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο της φιλοδοξίας που τρέφει προφανώς έτσι όπως έχει εκπεφραστεί αυτή η φιλοδοξία από πλευράς κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η στρατηγική αυτονομία σημαίνει ανεξαρτητοποίηση από κάποιον, αυτονομία εναντί κάποιου. Ε, στρατηγική αυτονομία σημαίνει να μπορεί κανείς να κάνει κάτι όταν οι άλλοι δεν θέλουν να το κάνουν και να έχει τα μέσα και τις δυνατότητες να εκπληρώσει την αποστολή που αποφασίζει να εφαρμόσει και να τρέξει. Σημαίνει Κανείς δεν είναι 100% αυτόνομος για να κάνει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μόνος του και δεν θέλει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γίνει συζήτηση και για τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ που είναι η βασική ε, ε, οργάνωση ασφαλείας και άμυνας στην Ευρώπη και έχει τεράστιες διαστάσεις και παρέχει συλλογική άμυνα και διάφορες, άλλε άλλες δηλαδή αποστολές εκπληρώνονται εντός ΝΑΤΟ. Πρέπει όμως να έχουμε τη στρατηγική αυτονομία, να τρέχουμε τις επιχειρήσεις που αποφασίζουμε να τρέξουμε. Ιδαλλιώς ούτε καν η διπλωματία και η πολιτική διάσταση δεν μπορεί να είναι λειτουργική εάν δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική αυτονομία. Εάν για παράδειγμα γίνεται λόγος να ε, έχουμε εμπάρκο όπλων στη θάλασσα, στη θαλάσσια οδό, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να το φροντίσει αυτό, να το περιφρουρήσει, να μπορεί να το εφαρμόσει και να έχει μέσα και εργαλεία και δυνατότητες ούτω ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτό το επίπεδο φιλοδοξία ότι θα αποκλείσει την ε, διακίνηση των όπλων διά τη ε, θαλάσσια οδού. Πρέπει να μπορεί να το ελέγξει αυτό. Άρα πρέπει να λύσει και το πρόβλημα του προϋπολογισμού. Αν βάλουμε όλες τις χώρες μαζί, είναι τεράστιος ο προϋπολογισμός, ο δεύτερος στον κόσμο, παγκοσμίω. Όποια αποστολή και αν ε, ε, θέλει κανείς να τρέξει, π.χ. μια εκπαιδευτική αποστολή, ανεξάρτητα αποστολή. Στρατηγική αυτονομία σημαίνει να μπορεί να την κάνει χωρί να ρωτήσει κανέναν. Αλλιώ δεν έχει αξιοπιστία. Δεν μπορεί να καθίσει στο τραπέζι και να ε, ε, καθίσταται αξιόπιστο εταίρο αν, αν δεν έχει αυτή τη στρατηγική αυτονομία. Επομένω, Τι σημαίνει στρατηγική αυτονομία αν το πάμε πολύ μακριά το πράγμα, ότι δηλαδή 27 χώρες θα μπορούν για, το, για ένα βασικό ζήτημα να μιλούν με μία φωνή. Στρατηγική αυτονομία επίσης σημαίνει ότι θα παρετηθεί κάποιος ελάχιστα κατά τη της ανεξαρτησίας του σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα και την ασφάλεια. Αλλά αυτό είναι σημαντικό γιατί θα δοθεί μεγαλύτερη εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τρέξει αυτές τις επιχειρήσεις. Και πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, είδε αλλιώς ε, χάνουμε ευκαιρίες. Και το 2011 είχε χαθεί πολλής χρόνος. Και πραγματικά, με κάθε ειλικρίνεια, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. There is no alternative. Αν δεν έχει κανείς τη στρατηγική αυτονομία να προτείνει μια επιχείρηση και πρέπει να πάει κάπου αλλού, να ζητήσει από κάποιον άλλο να μάθει, να ρωτήσει μήπως μπορείς εσύ να κάνεις την επιχείρηση αντί για μένα, ε, τότε, δεν, ε, τότε χάνει την αξιοπιστία του και δεν μπορεί ε, να ε, ισχύσει π.χ. στη Λιβύη ό,τι θέλουμε, την κατάπαυση της χρήση των στρατιωτικών μέσων, το εμπάργκο και το γιατί, γιατί ακριβώς δεν μπορεί αυτό να τα εφαρμόσει. για να το πω απλά. Μια χώρα ε, δεν έχει ένα στρατό για το ΝΑΤΟ, ένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα για τα Ηνωμένα Έθνη. Έχει ένα στράτευμα και αναλόγως με τις αποφάσεις ε, ε, παίρνει και την απόφαση που θα κατευθύνει αυτό το στράτευμα. Όταν όμως έχει στρατηγική αυτονομία, κάνει έρευνα και ανάπτυξη και φτιάχνει ένα καλύτερο στρατό και για την Ευρώπη, όπως βοηθάει περισσότερο και το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη και τους λοιπούς. Από εκεί και πέρα λοιπόν έρχεται μια στιγμή κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να παρέχει ισχυρά στρατεύματα στα Ηνωμένα Έθνη. Ήταν η περίπτωση του Λιβάνου πριν από τρία χρόνια. Τα περισσότερα στρατεύματα που αναπτύχθηκαν ε, ήταν ευρωπαϊκά και γίναμε αξιόπιστοι γιατί συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πράγματα που έχουμε δει και στο παρελθόν. Όταν κανείς αποφασίζει μια καινούργια αποστολή, γιατί έχει μια αυτόνομη βάση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προέρχεται και οφείλεται στη γεωπολιτική κατάσταση και τη γεωστρατηγική κατάσταση. Να μην επεκταθώ γιατί είναι περίπλοκο ε, το ζήτημα, αλλά Μάλλον το ΝΑΤΟ δεν θα ξαναπαίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα ε, μεγάλο ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με τα προβλήματα στη γειτονιά μας, όπως στη Λιβύη για παράδειγμα. Μιλούμε για συλλογική άμυνα, είναι ένας ε, τομέας που μας ενδιαφέρει κοινό τομέα γεωγραφικό που μα ενδιαφέρει, η Μέση Ανατολή, η Αφρική. Ε, η παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά σημαντική ε, εκεί. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε την ενοποιημένη ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μπορεί κανείς να καταβάλει πολύ σημαντικές διπλωματικές πολιτικές προσπάθειες και να αναπτύξει διάφορα εργαλεία και μέσα να αξιοποιήσει και να στηριχθεί από το στρατιωτικό σκέλος. Δεν υπάρχει μία και μόνη στρατηγική, στρατιωτική λύση, ειδικά σε δημοκρατικούς οργανισμούς. Σε πολλές αποστολές έχω δει ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση τα 40 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα ε, εάν ε, δεν έχει από πίσω το δυνατό, τη δυνατότητα να κινηθεί στρατιωτικά. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές δεν μπορεί κανείς να επιτύχει πολιτική ή διπλωματική λύση αν δεν έχει από πίσω να περιμένουν πλοία ε, πολεμικά ε, αεροπλάνα και ούτω καθεξής ε, έτσι ώστε να γίνεται αξιόπιστο. Το ίδιο ισχύει και για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη Σομαλία, το Μαλί. Όλη αυτή η περιοχή είναι εξαιρετικά σημαντική. Συνδέεται άρρηκτα με τη Λιβύη και με τα διάφορα σημεία που έχουν ξεσπάσει κρίσει στον κόσμο. Όπως είπα και στην παρέμβασή μου, αυτό που συμβαίνει στο Σαχέλ επηρεάζει τη Λιβύη και αυτό που συμβαίνει στη Λιβύη επηρεάζει το Σαχέλ. Είναι ένα συνδυασμό του φαινομένου ντόμινο με το φαινόμενο της πεταλούδας. με την ε, ε, πρέπει να γίνουμε ε, ρεαλιστές με την πτώση του χαλιφάτου πέφτουν τα πουλια του ντόμινο και επηρεάζουν και τις χώρες του Μαγκρέμπ και τις χώρες της Κεντρικής Αφρικής. Και αυτό είναι η βασική αποστολή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το capacity building, να εκπαιδεύσει και να ε, σφυριλατήσει το μηχανισμό ασφαλείας αυτών των χωρών για να μπορούν να λειτουργήσουν μόνες τους και να κάνουν τη δουλειά μόνες τους. Είναι όμως μεγάλο εγχείρημα αυτό γιατί δεν μπορεί κανείς να φτιάξει στρατό εκ του μηδενός, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται μέσα, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται συμβουλευτική και ούτω καθεξής. Τώρα με το EUTM με την εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Training Mission, πρέπει να αποκτήσει πιο μεγάλα φτερά, πρέπει να γίνει πιο δυνατή. Δεν είναι το θέμα η εκπαίδευση, είναι το θέμα η δημιουργία ικανοτήτων χωρών. Πρέπει κανείς να είναι χορηγός, να, είναι, ε, να τους πλαισιώνει, να τους βοηθά τις χώρες αυτές. Είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός αυτή τη στιγμή. Και ε, δεν είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν πιο ισχυρές αυτές οι δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν είναι ιδιαίτερα παρούσες στο εξωτερικό. Ό,τι και να σας πούν, ό,τι και να ακούσετε, μην το πιστεύετε. Πριν από 10 χρόνια είχαμε πέντε φορές περισσότερες δυνάμεις στο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεπτυγμένες. Όμως οι αποστολές μας δεν είναι αρκετά αξιόπιστες, ε, ε, δεν γίνονται αντιληπτέ ως αρκετά αξιόπιστες από τα κράτη-μέλη. Είναι μικρές, δεν ασκούν μεγάλη επιρροή γιατί το μόνο που κάνουν είναι εκπαίδευση. Άρα, αν μπορέσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας και η εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, εμπλουτιστεί, να μην δίνει μόνο εκπαίδευση αυτή καθεαυτή, αλλά να κάνει συμβουλευτική και αν διασφαλίσουμε την προστασία αυτών των δυνάμεων, γιατί δεν εμπλέκονται σε μάχη, τότε θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία, γιατί οι εκπαιδευτικές αυτές αποστολές λαμβάνουν χώρα στις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου και αν κανείς κάνει εκπαίδευση υπάρχει το ενδεχόμενο να τον πυροβολήσει κάποιος σε μια ε, επικίνδυνη περιοχή στη Σομαλία. Ε, το να διασχίσει κανείς το Μογκαντήσου για να πάει να κάνει εκπαίδευση είναι σαν να διασχίσει την πιο επικίνδυνη περιοχή του Αφγανιστάν και άρα μπορεί να υποστεί πειρά. Είναι πολύ δυστυχές το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να καταλάβει ότι το ένα πράγμα χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση, περιφερειοποίηση, επιπρόσθετες δυνάμεις. Και οπωσδήποτε η ιδέα ε, του να ενδυναμωθεί όλη η διαδικασία είναι θέμα προστασίας κιόλας ε, και οπωσδήποτε θα πρέπει η αποστολή να είναι ασφαλής, θα πρέπει ο διοικητής να έχει ε, όλες τις δυνατότητες διοίκησης από εκεί και πέρα βεβαίως η κάθε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στην αποστολή είτε είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία ε, θα έχουν την ε, δυνατότητα να ε, συζητήσουν τα θέματα αυτά. Υπάρχουν αποστολές οι οποίες υποστηρίζονται περισσότερο από μία χώρα και λιγότερο από τις υπόλοιπες κτλ. Και στο Μαλί αλλά και αλλού έχουμε πέντε αποστολές. Στο Μαλί είναι πέντε οι αποστολές Έχουμε κοινή αποστολή, έχουμε ε, γαλλική αποστολή, ε, την UTM, ε, έχουμε την αποστολή του, του Σαχέλ και έχουμε και τις, το συντονισμό των τοπικών δυνάμεων και έχουμε και τη δυνατότητα παροχής ε, κατάρτισης ε, ε, και βεβαίως αυτή η ιδέα για την προστασία του στα είναι μια πολύ καλή ιδέα, τρομερή ιδέα, αλλά είναι ακόμα ιδέα. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα εργαλεία τα οποία θα υποστηρίξουν αυτές τις ιδέες διαφορετικά. Θα συνεχίσουμε να έχουμε αποτυχημένη κατά κάποιο τρόπο προσπάθεια το Σαχέλ δεν πρόκειται να ε, ε, σωθεί από μόνο του, δεν πρόκειται να υποστηριχθεί από μόνο του. Πολλά Πολλές είναι ε, οι περιπτώσεις στην Αφρική όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβουμε ευθύνη ή να συνεχίσουμε την ανάληψη ευθύνη που έχουμε πάρει. Okay, we can put the European Facility in this just because it's important. Ναι, το θέμα του Ταμείου, του ε- Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου, ε, πρέπει να είναι απλό, πρέπει να είναι αποτελεσματικό, να έχει τη δυνατότητα ε, γρήγορης προσέγγισης ε, και αντιμετώπισης, δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν εταίροι, διαδικασίες εκπαιδευτικές και άλλες, δυνατότητα να παραχθούν assets από πλευράς των κρατών μελών Ε, συνήθως τις αποστολές ε, το Ηνωμένα Έθνη πληρώνουν ε, για τους στρατιώτες και το μείγμα τα υπόλοιπα. αλλά υπάρχει και η συντήρηση, υπάρχει η ο εξοπλισμός που παρέχουμε ας πούμε στο Μαλί, το πετρέλαιο για να κινούνται τα οχήματα κτλ. Και έχουμε αυτή την υποστήριξη. Εμείς δεν υποστηρίζουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αυτές τις αποστολές. Το αμυντικό ταμείο λοιπόν τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, κεντρικής σημασίας. Ε, χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για την έρευνα και την ε, ανάπτυξη. Ανάπτυξη είτε πρόκειται για ε, αμυντικά συστήματα είτε για άλλα ε, θέματα Ε, ας πούμε, τι να σας πω, έχουν, έχει χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 7 θωρακισμένων, μετά δεν έχουμε όμως αναβαθμίσεις ε, και στην ουσία μετά από λίγο χάνονται τα χρήματα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε πιο αποτελεσματικά εργαλεία. Στην Military Committee διαπιστώνουμε συχνά ότι υπάρχουν assets ε, που έχουμε στην διάθεσή μας, αλλά ε, δεν είναι εύκολο να δοθούν από τον ένα στον άλλον. Πρέπει να διευκολυνθούν οι διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος συντονισμός. ενδεχομένως δηλαδή να υπάρχει ένα κοινό ε, ε, οπλικό σύστημα και η κάθε χώρα να συμμετέχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ε, ή ή σε κάθε περίπτωση διαγωνισμού η κάθε χώρα να βάζει συγκεκριμένο οικονομικό. Εμείς ε, προωθούμε την σκέψη όσον αφορά διάφορα στρατιωτικά ε, σενάρια ή εναλλακτικές ε, λύσεις. Ε, βεβαίως το θέμα είναι να έχουμε ε, ακριβώς ε, και στα πλαίσια της ΕΟΦΟΡ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλες τις απειλές. Εν πάση περιπτώσει αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει στερεωτική παρουσία από όλες τις χώρες που θα δουλέψει όσο γίνεται καλύτερα και θα επενδυθούν επομένω ε, οι πόροι που θα δαπανηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέραν αυτού βεβαίω ε, οι πολιτικοί θα αποφασίσουν, είναι πολιτικού επίπεδου η απόφαση. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται πριν από την πολιτική απόφαση. Το ίδιο ισχύει και με το EDF, με το ε, Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Είναι σημαντικό να δώσουμε εμείς, να παράσχουμε εμείς ε, την ε, δικιά μας ε, στρατιωτική συμβουλή και προς τη βιομηχανία και προς Εμείς Ευελπιστούμε ότι ε, θα ε, προχωρήσει η διαδικασία. Ο πρόεδρος της ε, Military, ως πρόεδρος της Military Committee, εγώ θέλω να εμπλέκομαι με τις διαδικασίες του Αμυντικού Ταμείου και θεωρούμε ότι όλα θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε ο τελικός χρήστης να έχει τη σωστή πληροφόρηση ε, και ε, εν τέλει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση ε, των πόρων που έχουν εμπλεκεί σε όποια διαδικασία. Το θέμα της μετανάστευσης τώρα. Δεν αναφέρθηκα με την πολιτική, το πολιτικό σκέλος του, της μετανάστευσης, αλλά με το τεχνικό. Για να λυθεί το πρόβλημα, όντως θα πρέπει να πάμε να βρούμε τις ρίζες του προβλήματος. Ε, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει τρομοκρατία, ε, υπάρχουν ε, διάφορες ε, κρίσεις διαφόρων ειδών δηλαδή. Αυτά είναι τα αίτια της μετανάστευσης. Δεν είναι δυνατόν να απομονώσουμε ένα από όλα αυτά τα προβλήματα. Ε, δηλαδή έχουμε τρομοκρατία, μετανάστευση από, από συντονισμό ε, και θα πρέπει να έχουμε μία γενικευτική προσέγγιση έτσι ώστε να λύσουμε το ευρύτερο ε, πρόβλημα. Ε, ενδεχομένως χάσαμε μια γενικευτικη προσεγγιση ετσι ωστε να λυσουμε το ευρυτερο προβλημα ε ενδεχομενως χασαμε μια ευκαιρια στην ε, Λιβύη. Η Λιβύη ξεκίνησε ήδη από το 2011, τώρα είμαστε 2020. Έχουν μεσολαβήσει 9 χρόνια, σειρά και των οποίων η Ευρώπη θα έπρεπε ίσως να έχει βρει μια ενιαία φωνή και τη δυνατότητα να κάνει κάτι πιο συγκεκριμένο. Τώρα είναι αργά, αλλά όχι υπερβολικά αργά. Ε, όπως ε, και την τελευταία στιγμή δεν ήταν, αρκετά, δεν ήταν υπερβολικά αργά έτσι ώστε να κερδίσουμε ε, τον πόλεμο κατά των Ναζί, έτσι ε, και τώρα έχουμε ακόμα χρόνο. Η Σοφία είναι η μόνη αποστολή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και που συνδέει την Ευρώπη με την Νότια Μεσόγειο και την Λιβύα. Χρειάζεται βέβαια, χρειάζονται πόροι, χρειάζεται συμφωνία από όλες τις πλευρές. Ε, και ε, είτε ε, πρέπει να το δουλέψουμε και μέσω του Συμβουλίου. Η Σοφία δεν θέλει να σώζει μετανάστες. Δεν είναι αυτός ο πρώτος της στόχος. Είναι να καταρτίζει, να εκπαιδεύει τους, την ακτοφυλακή των ε, άλλων χωρών, αλλά βεβαίως ε, τα πλοία μας ε, και οι κυβερνήτες μας πάντα έχουν την ηθική υποχρέωση να σώζουν ζωές. Και ούτως ή άλλως, ακόμα και σε μεσούντος πολέμου, η ηθική υποχρέωση, και αυτό κάνουν όλοι οι διοικητές, είναι να σώζουν ζωές. Εγώ ως στρατιωτικός λέω ότι το γεγονός ότι κινούμαστε γρήγορα και σωστά έτσι ώστε να καλύπτουμε κενά, αυτό ε, είναι πιο σοβαρό από τον αριθμό των ε, μεταναστών που μπορεί να ε, σώσουμε ή που μπορεί μετά να επαναπροωθηθούν κτλ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 700.000 μετανάστες ε, στην ε, Λιβύη που ενδεχομένως εάν λυθούν κάποια προβλήματα θα φύγουν ε, από τη χώρα. Ναι, χρειάζεται καθοδήγηση, πρέπει να επιμείνουμε στο εμπάργκο των όπλων και θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτήν την επιχείρηση η οποία είναι η μόνη που υφίσταται ακόμα. υποστηρίζω λοιπόν στεναρότατα την επιχείρηση Σοφία. Ε, η γενική της ε, αρχή είναι μια ε, σωστή αρχή και βεβαίως το θέμα των αποβάσεων στα λιμάνια δεν είναι στρατιωτικό ζήτημα. και το σημαντικό είναι να ε, καταφέρουν οι 27 να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ασφάλειας, μια κατάσταση ε, ασφάλειας ε, και βεβαίως μετά μπορεί να υπάρξουν και άλλες επιχειρήσεις ή αποφάσεις παύσης πυρός κλπ. Ευρώπη και ΝΑΤΟ, βεβαίως εμείς θέλουμε συνεργασία. Άλλωστε αναφέρεται και στις αρχές της Global Strategy. όχι γιατί ε, οι περισσότεροι από τους 27 είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά ε, και γιατί γενικότερα χρειαζόμαστε μια ισχυρή συνεργασία. Ο συντονισμός είναι αρκετά περιορισμένος προς ώρας και ε, αυτή την ώρα διέπονται οι σχέσεις από το ε, ε, Berlin Plus, ωστόσο μπορεί να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση επίλυση σε κάποιων προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό θα πρέπει συγκεκριμένα κρατημέλη να το αποφασίσουν. Και μετά να βρεθούν οι τεχνικές ας πούμε ε, δυνατότητες, ε, καταρτήσεις, εκπαιδεύσεις κλπ. Αλλά ξέρετε, εντό στρατηγική αυτονομία ε, κάτι τέτοιο θα γίνει υποχρεωτικό γιατί με το Berlin Plus έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη δομή του ΝΑΤΟ για τι επιχειρήσεις του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρησιμοποιούμε το NATO Command για την ώρα, ε, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα γενικά. Thank Αυτά ήθελα να σας πω. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ, ε, στρατηγέ, για αυτές τις πολύ σαφείς απαντήσεις που μας δώσατε. Ε, και εμείς προβληματιζόμαστε με τους δικούς σας προβληματισμούς. σημεριζόμαστε λοιπόν τους προβληματισμούς σας. Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα και θέλω να καλωσορίσω τον Καμίγ Γκόν και την Αλεξάνδρα διευθύντρια ε, ε, του γραφείου του German Marshall Fund στο Παρίσι για να ε, έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 70η επέτειο του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο αρκετά τεταμένη και με αρκετέ αλλαγέ. Η Βορειοατλαντική ε, Συμμαχία χρειάστηκε να προσαρμόζεται στι νέε προκλήσει ασφάλεια και άμυνα καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργία τη, αρκεί να αναφέρουμε την τρομοκρατία μετά τι 11 Σεπτεμβρίου 2001, που οδήγησε στην πρώτη ενεργοποίηση του άρθρου 5 τη συνθήκη τη Washington E την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών. Και πιο πρόσφατα, 3 και 4 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο, οι επικεφαλής κάθε χώρας του ΝΑΤΟ αποφάσισαν να αναγνωρίσουν το διάστημα ως νέα διάσταση ε, άμυνας και να ξεκινήσει ένας προβληματισμός για το μέλλον του ΝΑΤΟ και για τους στόχους του γιατί είναι αναντήρητο ότι το θέμα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του ΝΑΤΟ τίθεται οξύτατα στο διεθνές πλαίσιο αυτή τη στιγμή με μία επάνωδο σε μονομερείς ε, αποφάσεις, με ένα ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων και με μία επανεφάνιση εθνικισμών. Και ενδεχομένως ε, και κάποιες ερωτήσεις για την έννοια της λέξης «συμμαχία». Η διάσκεψη του ΝΑΤΟ δεν ήταν κάτι που θα φοβόμασταν ότι απλώς προσπαθούσαν ε, οι συμμετέχοντες να τηρήσουν τις δημοσιονομικές τους δεσμεύσεις. Δεν ήταν καθαρά λογιστικό το αποτέλεσμα, αλλά μπόρεσε να τεθεί σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης σύγκλησης και στρατηγικών προσανατολισμών. Η διακήρυξη που εγκρίθηκε στο Λονδίνο, που υπάρχει στο φακελό σα, υπενθυμίζει ότι η ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ εταίρων, ε, όπως το άρθρο 5 και η συνοχή είναι βασικές αρχές της συμμαχία δεν πρόκειται μόνο για μια σημασιολογική διαφορά μεταξύ του να είμαστε ε, ε, σύμμαχοι ή όχι. Καμία χώρα της συμμαχίας δεν μπορεί να μην επηρεάζεται από αποφάσεις άλλων, ιδίως όταν υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια κάθε κράτους. Οι πρόσφατες επιλογές της Τουρκίας βεβαίως και θέτουν οξύτατα ζητήματα για την λειτουργία της συμμαχίας και είναι απαραίτητο να συζητήσουμε και το πεδίο δράσης του ΝΑΤΟ σε ολόκληρο τον κόσμο τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να συμμετάσχει η συμμαχία περισσότερο στη Μέση Ανατολή χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη επακριβώς ποια είναι η σημασία μιας τέτοιας προσδοκίας και αν η σημασία αυτού του θέματος θα μπορούσε ε, να σημαίνει μεγαλύτερη αποδέσμευση των αμερικανικών στρατευμάτων. Όλα αυτά εντάσσονται και στο πλαίσιο πρωτοβουλειών για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων άμυνας και ε, της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Στο Λονδίνο, πολύ σωστά χαιρετίστηκαν ε, οι άνευ προηγουμένου πρόοδοι αυτής της συνεργασίας. Θέλουμε η υποεπιτροπή μας να συμμετάσχει στον προδιορισμό των ε, κοινών ε, θέσεων για την ασφάλεια και την άμυνα και στην ενίσχυση ε, τη συνεργασία μας, ιδίως διατηρώντας στενή συνεργασία και διάλογο με τις, με του ΝΑΤΟ. Θέλω να δώσω το λόγο στην Αλεξάνδρα Ντεχόπ Σέφερ για λίγα λεπτά και μετά στον Καμίγι και μετά να ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ Ναταλή Λουατζό, ευχαριστώ όλους ε, τους παρόντες σήμερα εδώ. Για μένα είναι ε, τιμή και χαρά το ότι βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να συζητήσουμε για το ΝΑΤΟ σε μια περίοδο που ε, ε, είναι πολύ σημαντική για το ΝΑΤΟ. Και θέλω τώρα να μιλήσω αγγλικά, αλλά όλοι σας είστε είτε δήλωση είτε τρίγλωση εδώ, άρα είμαι σίγουρη ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Όπως είπε η Ναταλή, είμαι διευθυντρία του Γερμανικού Ταμείου Μάρσαλ στο Παρίσι, επομένως ε, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε σήμερα είναι να έχουμε ευρωπαϊκή αλλά και διατλαντική συζήτηση για τα θέματα τα οποία τίθενται για τους Ευρωπαίους και για τους Αμερικανούς συμμάχους. Όταν ε, μιλάμε για το ΝΑΤΟ, πάντοτε θέλω να αναφέρομαι σε κάτι που ίσως έχετε ήδη διαβάσει το έργο του Steve ε, Watts Peace ε, που είχε δημοσιευθεί σε ένα περιοδικό γιατί οι συμμαχίες ε, παραμένουν ή καταραίουν. Αυτός είναι ο τίτλος εκείνου του άρθρου. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό το άρθρο. Τα βασικά επιχειρήματα που είχε αναφέρει τότε συνοπτικά έλεγαν ότι αυτό που συζητάμε σήμερα είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι η κοινότητα συμφερόντων και η δεύτερη είναι η κοινότητα αξιών που είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες και όταν ο ένας πυλώνας γίνεται ευάλωτος γίνεται και ο άλλος πυλώνας ευάλωτος. Θα ήθελα να σας αναφέρω τέσσερα βασικά ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια οποιαδήποτε σοβαρή ανάλυση για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Το ένα είναι η μεταβαλλόμενη έννοια της απειλής, το δεύτερο η πιθανότητα, το τρίτο η πολιτική ηγεσία και η επιρροή των εσωτερικών πολιτικών μας, των εγχώριων πολιτικών μας, ε, στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της συμμαχίας και το τέταρτο που ανέφερε και η Ναταλή για η Ευρώπη και πώς η Ευρώπη μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικός πυλώνας ασφάλειας και πώς μπορούμε να ενισχύουμε αυτή τη διατλαντική σχέση. Το πρώτο λοιπόν θέμα που έχει άμεση σχέση και με την αλληλεγγύη, ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με την ανατολική, νότια πτέρυγα. Δεν μου αρέσουν αυτού του είδους τα σύνορα μεταξύ ε, ε, είναι λίγο τεχνητές αυτές ε, οι έννοιες. Αν δούμε το ρόλο του ΝΑΤΟ και στα δύο αυτά μέτωπα, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι χρήσιμο να συζητάμε την έννοια της απειλής μέσα στην συμμαχία. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι πώς μια συμμαχία τον 21ο αιώνα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Είμαστε στο μέσο όλων αυτών, αυτού του, προβληματισμού. Ανέφερε και η Νατέλη τι σημαίνει το να είμαστε μια συμμαχία, τι σημαίνει το να είμαστε σύμμαχοι. Μια συμμαχία είναι μια εξελισσόμενη έννοια. Έχει σχέση με τη γεωπολιτική, με απειλές που εμφανίζονται ή εξαφανίζονται και αν δείτε τις στρατηγικές έννοιες ε, το 91 τέλος του ψυχρού πολέμου, το 99 μέσα του πολέμου στο Κωσυφοπαίδιο και 2010 στο μέσο του πολέμου στο Αφγανιστάν βλέπετε ότι οι στρατηγικές έννοιες, η στρατηγική διαδικασία της συμμαχίας καθοδηγείται από τις κρίσεις, από τη βάση προς τα πάνω και κατά πολύ από τις προτεραιότητες των ΗΠΑ. Γι' αυτό όταν ο πρόεδρος λέει η Αμερική πάνω απ' όλα ή ε, ε, ότι το ΝΑΤΟ είναι ευρωπαϊκή οργάνωση, εν πολύ στην αμερικανική οργάνωση ε, το ΝΑΤΟ και πρέπει να δούμε πώς μπορεί το ΝΑΤΟ να παίζει ένα πιο σφαιρικό ρόλο για την τεχνολογία, για το διάστημα, για ζητήματα που έχουν σχέση με την Κίνα, ενίσχυση του ρόλου του έναντι της τρομοκρατίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα που σαφώς ε, συμβαδίζουν με τα αμερικανικά συμφέροντα. Κάτι που θέλω να τονίσω είναι ότι μετά ε, την 11η Σεπτεμβρίου και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί σύμμαχοι υπέπεσαν ε, σε μια στρατηγική παράλυση για τον, με τον παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και ακόμη λειτουργούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και ο Γενικός ε, Γραμματέας του ΝΑΤΟ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχτές αυτό τόνισε η υπαριθμόν ένα αποστολή του ΝΑΤΟ της Διατλαντικής ε, Συμμαχίας είναι η τρομοκρατία, η Ρωσία και η Κίνα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι αυτό μας έχει εμποδίσει από ένα ευρύτερο προβληματισμό σε ένα ευρύτερο στρατηγικό περιβάλλον. Ξαφνικά ανακαλύψαμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι η Κίνα ανέρχεται πάρα πολύ γρήγορα, ότι η Ρωσία ε, είναι σαφώς ένας παράγων και στη δική μας περιοχή. Όλα αυτά είναι γεωπολιτικές και στρατηγικές προκλήσεις. Πρέπει λοιπόν, πιστεύω, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μας προβληματίσουν αυτές οι βαθύτερες τάσεις που επιταχύνουν αυτά με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Και πρέπει να δούμε αυτό ε, το νόημα του στρατηγικού πλαισίου. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που ήθελα να σας αναφέρω. Το δεύτερο αφορά ε, τη μετεξέλιξη του θεματολογίου του ΝΑΤΟ και των προτεραιοτήτων. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις μετά από την, ε, τις δηλώσεις Τραμπ ε, για το ΝΑΤΟ και όλα αυτά έχουν σχέση με την αποστολή ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση να εμβαθύνει τη δέσμευσή του στη Μέση Ανατολή το ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μίλησε για πρόληψη μάλλον παρά για παρέμβαση. Είμαστε σε μια στρατηγική προσπάθεια ελέγχου ελέγχου της τρομοκρατίας, ελέγχου των ροών μετανάστευσης και περιφερειακά και τοπικά στο μέτρο του δυνατούν. Και παράλληλα, το ΝΑΤΟ παραμένει στρατηγική συμμαχία και το πρωταρχικό εργαλείο είναι το στρατιωτικό εργαλείο και δεν είναι προσαρμοσμένο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με αποτυχημένα κράτη, με την τρομοκρατία, με όλα αυτά που χρειάζονται περισσότερο υβριδικά εργαλεία. Και θα πρέπει σε αυτά να συνεργάζονται πολύ περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αλλά υπό την Αμερικανική έννοια, οι ιδέες του Πενταγώνου αυτή τη στιγμή επανεξετάζονται. Προσπαθεί το Πεντάγωνο να επανεξετάσει το ίχνος του παντού, στην Αφρική, στην Μέση Ανατολή. Προσπαθούν να δουν πώς μπορεί το ΝΑΤΟ να αναλάβει δράση σε τομείς όπου θέλουν να, θέλουν να αποσυρθούν οι ΙΠΑ. Και αυτό έχει άμεσα σχέση ε, με το θέμα που έθεσε ο Τραμπ για το ΝΑΤΟ και τη ΥΠΑ. Και το Σαχέλ είναι όντως ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα διότι το Πεντάγωνο τέλος Ιανουαρίου θα ε, υποβάλει σχέδια μερικής αποχώρησης. Αυτό έχει επιπτώσεις και για μας, κυρίως για τη Γαλλία στο Σαχέλ, αλλά και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί θυμάμαι ότι ήμουν στο Κέντο ήμουν στο προσωπικό πολιτικής ασφαλείας ε, όταν συζητούσαμε τα θέματα της, ε, των επιχειρήσεων στη Λιβύη το 2011. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ήθελαν να το επαναθέσουν στο ΝΑΤΟ και μου φάνηκε περίεργο, σαν να μην ήταν η ΙΠΑ κομμάτι του ΝΑΤΟ, σαν το ΝΑΤΟ να ήταν ευρωπαϊκή οργάνωση. Και έχω και τώρα ε, το ίδιο αίσθημα με τη Συρία, το Ιράκ, ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει το ρόλο του. Δεν είναι ε, μεταφορά ε, του βάρους, ε, πρέπει να είναι επιμερισμός των βαρών. Και γι' αυτό χρειάζεται να γίνει μια τέτοια συζήτηση με τους Αμερικανούς συμπάχων μας για το πώς καταμερίζονται τα βάρη. Το δεύτερο σημείο, η αξιοπιστία, όντως πιστεύω ότι ο στρατιωτικός και ο πολιτικός πυλώνας απομακρύνονται μέσα στο ΝΑΤΟ. Και η παρέμβαση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία ε, το αποκάλυψε αυτό, χωρίς διαβούλευση έγινε. Από το 2013 τίθεται το θέμα αυτό ε, στη Γαλλία και ενισχύθηκε με τον Τραμπ. Πόσο μπορούμε να βασιζόμαστε στους Αμερικανούς συμμάχους μας. Και όταν αρχίζουμε να θέτουμε τέτοια ερωτήματα, σημαίνει ότι η θεμελιώδης αρχή του ΝΑΤΟ, η εμπιστοσύνη, αμφισβητείται. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Δεν είναι πρώτη φορά που θέτουμε το ερώτημα αυτό που διαρωτώμαθα κατά πόσο χρειάζεται περισσότερη πολιτική διαβούλευση. Αν θυμηθείτε την κρίση του Σουέζ το 1956, την Επιτροπή των Τριών, Νορβηγία, Ιταλία, Καναδάς, τόνιζε την ανάγκη για μεγαλύτερη πολιτική διαβούλευση. Έκθεση Harvard το 1974 που τόνιζε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του στρατιωτικού και του πολιτικού πυλώνα και αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί και μάλιστα με κάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει ακόμη, δηλαδή μια επαναξιολόγηση των τελευταίων στρατιωτικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση, να καταγράψουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων στρατιωτικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ από την 11η Σεπτεμβρίου παραδείγματος χάρη, τι έχει πάει στραβά, τι μπορούμε να διορθώσουμε. Θέλω να κάνω μια σύντομη σύγκριση. Πριν από 15-20 χρόνια αυτό που, που αποκαλούσαμε παρέμβαση βασιζόταν σε κάποιες υποθέσεις. Πρώτον ότι η ΕΠΑ είναι εγγυητής της παγκόσμιας τάξης. Δεύτερον η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό των ΗΠΑ. Και τρίτον δεν υπήρχαν ε, κάποιοι σοβαροί παράγοντες που να αμφισβητούν την κυριαρχία των ΗΠΑ στη Δύση. Αν όλα αυτά τα δείτε στο σημερινό πλαίσιο, είναι πολύ διαφορετική εικόνα. Ε, καταρχήν, οι ΕΠΑ ε, αποχωρούν από αυτό που θεωρεί, θεωρεί, θεωρεί το ε, υπευθυνότητα των ΗΠΑ. Δεύτερον, η Ευρώπη είναι διερημένη, ιδίω αν δείτε θέματα όπως η Λιβύη και άλλα. Και τρίτον, υπάρχουν κάποιες αυταρχικές δυνάμεις που παρεμβαίνουν όλο και περισσότερο που επωφελούνται από τις διαιρέσεις στο, δικό, στο εσωτερικό το δικό μας. Επομένως, βρισκόμαστε σε μία στιγμή που πρέπει να εξετάσουμε την έλλειψη πολιτικής συνοχής και να προσπαθήσουμε να το επανεξετάσουμε, γιατί αυτό έχει επιπτώσεις στην αξιοπιστία μας και στην εμπιστοσύνη μέσα στη συμμαχία. Τρίτον, η ηγετική σχέση. η ηγετική θέση των ΗΠΑ παραμένει ιδιαίτερα παρούσα μέσα στο ΝΑΤΟ. Η ιδέα του ΝΑΤΟ που ε, υπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ παγκοσμίω. Σε αυτό έχουμε επανέλθει. Και αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας μας, γιατί έχουμε αυξήσει τον προπολογισμό της άμυνας, έχουμε δείξει τη χρησιμότητά μας και τώρα η κυβέρνηση Τραμπ ε, δρέπει τα ωφέλη του ΝΑΤΟ, που μπορεί να είναι εν μέρη καλό και εν μέρη μη καλό, διότι ο Τραμπ προσπαθεί να καθοδηγήσει το θεματολόγιο του ΝΑΤΟ. Και δεν πιστεύω καθόλου στην συζήτηση του ότι μπορεί να αποχωρήσουν οι ΙΠΑ από το ΝΑΤΟ. Αντιθέτως πιστεύω ότι οι ΙΠΑ θα συνεχίσουν να ηγούνται του ΝΑΤΟ, θα συνεχίσουν να επενδύουν στο ΝΑΤΟ και θα συνεχίσουν ε, να είναι όλο και περισσότερο απαιτητικοί έναντι ημών των Ευρωπαίων εταίρων για τον απλούστατο λόγο ότι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με την Κίνα το ΝΑΤΟ η Ουάσιγκτον το βλέπει ως σημαντικό στρατηγικό κυματοθράφστη, ιδίως για να κρατήσει την ηγεμονία των ΗΠΑ στην αμυντική αγορά της Ευρώπης. Αναφύεται λοιπόν μια ευκαιρία, μια διατλαντική ευκαιρία για να παραμείνουν οι ΗΠΑ αξιόπιστοι εταίροι μέσα στο ΝΑΤΟ, μειώνοντα τη στρατιωτική τους ε, συμμετοχή και σε αντάλλαγμα από τους Ευρωπαίους θα ζητηθεί να περιορίσουν ε, την είσοδο των Κινέζων ε, σε προηγμένες τεχνολογίες και σε στρατιωτικά προϊόντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά αναδύεται με έναν σταδιακό αλλά συνεχή τρόπο μετά το 2020 και την εκλογική εξατία στη ΣΥΠΑ δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν αυτά. Μπορεί να ακολουθήσουν μια πιο διπλωματική γλώσσα, αλλά το θέμα της κατανομής των βαρών, το 2% η προτεραιότητα στην Κίνα, η Ευρώπη που φαίνεται ως ε, ε, χρηστικό ε, εργαλείο σε αυτό τον το παγκόσμιο ανταγωνισμό με την Κίνα, αυτά θα παραμείνουν. Βλέπω κυρίως τη γαλλική θέση από τη θέση μου στη Γαλλία και βλέπω ε, ποιες είναι οι τάσεις και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω και για την ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να εμβαθύνουμε αυτές τις ε, ε, σχέσεις Μιλάμε για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε και ξέρω ότι είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα προκλητικά να αναφέρω ότι αυτό είναι κάτι που ήδη κάνουμε, δηλαδή ε, δρούμε στρατηγικά σε πολλ... με πολλούς τρόπους, διπλωματικά στο Ιράν, μη αποδεχόμενη την απόφαση των ΗΠΑ, παρότι εξαναγκαστήκαμε σε κάποιο βαθμό να προσεγγίσουμε τη θέση των ΗΠΑ, στο θέμα του κλίματος δεν ακολουθούμε ε, τις ΙΠΑ σε αυτό το θέμα. Θαλάσσια ασφάλεια, αν δείτε στα στενά του Ορμούς. όλα αυτά είναι θέματα όπου ήδη την Ευρώπη τη βλέπουμε περισσότερο στρατηγικά αυτόνομη, διπλωματικά, επιχειρησιακά περισσότερο αυτόνομη σε σύγκριση με τις αποφάσεις των ΗΠΑ. Και είναι μια υγιής στάση αυτή πιστεύω. Αυτό το οποίο μας διαιρεί στο εσωτερικό της Ευρώπης και στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσελ, προσπαθούμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων Αμερικανών και Ευρωπαίων για να δούμε προς τα που κινούνται οι ΙΠΑ και οι διατλαντικές σχέσεις και δεν έχουμε πάντοτε την ίδια εικόνα όλοι οι Ευρωπαίοι για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων. Και αυτό φαίνεται και από τη συζήτηση που κάνουμε για το τι σημαίνει στρατηγική αυτονομία. Υπάρχουν οι σκανδιναβικέ χώρες της Βαλτικής που βλέπουν τη στρατηγική αυτονομία ως κάτι που αποδυναμώνει τις διατλαντικές σχέσεις. Η Γαλλία έχει μια κάπως μοναδική σχέση που λέει αντιθέτως. Θα είμαστε καλύτεροι εταίροι για τη ΣΥΠΑ με τη στρατηγική αυτονομία και κάπου στο μέσο βρίσκεται η Γερμανία και η Βρετανία που λένε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε περισσότερο ανεξάρτητα και μου έκανε εντύπωση ο Υπουργό Άμυνα ε, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσφατα, που είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να σκέφτεται πιο ανεξάρτητα από τι Ηνωμένε Πολιτείε στο μέλλον για τι διάφορε συγκρούσει, ε, θέτοντα σε προτεραιότητα το πλαίσιο του ΝΑΤΟ πάντοτε. Και κλείνοντα, θα ήθελα να πω τα εξή. Αντί να εστιάζουμε στο αν θα πρέπει να έχουμε στρατηγική αυτονομία, αν οι ΕΠΑ θα πρέπει ε, να έχουν μεγαλύτερη δέσμευση ευρωπαϊκή, στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου τα ευρωπαϊκά συμφέροντα για θέματα ασφάλειας. Πώς θέλουμε να είμαστε σημαντικός παράγων σε αυτό τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ ΕΠΑ και Κίνας. Και ε, έχω τρεις προτάσεις. Πιστεύω ότι το μέλλον της Ευρώπης ε, ως παράγοντος ασφαλείας και η μελλοντική ισχύ της Διατλαντικής Συμμαχίας εξατάται από το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη κατά τρία διαφορετικά σημεία. Πρώτον, με τη ΣΥΠΑ, κατά πολέμηση της τρομοκρατίας, η Κίνα είναι ένας τομέας όπου πρέπει να ενισχύσουμε τη Διατλαντική Συμμαχία. Δεύτερον, χωρίς τις Ηνωμένε Πολιτείε και όπως σας είπα ήδη αυτό το κάνουμε με πολλές εκφάνσεις και η στρατηγική αυτονομία ακριβώς αυτό δείχνει αυτή η συζήτηση. Και το τρίτον, μαζί με άλλες δυνάμεις, διότι μερικές φορές ομφαλοσκοπούμε και πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε τον κόσμο σήμερα όπως είναι πραγματικά. Βλέπουμε μια νέα γεωπολιτική εποχή. Η Διατλαντική Συμμαχία δεν αρκεί πάντοτε όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και βεβαίως και πρέπει να συνεργαζόμαστε και την ε, εταιρική μας σχέση να τη σκεφτόμαστε ευρύτερα και ίσως με πιο πολύπλοκους εταίρους όπως η Ρωσία, η Τουρκία και άλλοι. Δεν είναι λοιπόν απεσιόδοξη η εικόνα που έχω για τη Διατλαντική Συμμαχία τα επόμενα χρόνια. Αρχίζει περισσότερο ε, μία τμηματική αντιμετώπιση, δηλαδή συνεργαζόμαστε σε τομείς όπου έχουμε κοινά συμφέροντα και σε άλλους τομείς θα πρέπει να σκεφτόμαστε ως Ευρωπαίοι περισσότερο αυτόνομα και άλλοι τομείς όπου θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με άλλους εταίρους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ίσως μακρηγορήσατε κάπως και θα πρέπει και οι συνάδελφοι να μπορούν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Γκραντ έχει το λόγο αυτή τη στιγμή. Έχω την ευχέρεια, είμαι στην ευχάριστη θέση κυρία Πρόεδρε, να μιλήσω δεύτερος. Και η προηγούμενη ομιλήτρια, η Αλεξάνδρα Ντεχούπ Σέφερ, ήδη κάλυψε πολλά ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το στρατηγικό περιβάλλον. Και άρα δεν χρειάζεται να χρονοτριβήσω. Επίση, στο αφεντικό μου, ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ήταν ενώπιον τη Σχετική Επιτροπή πριν από δύο μέρε και άρα έχει ενημερώσει το Κοινοβούλιο για το όραμά μας, για την ε, γενικότερη επισκόπηση που κάνουμε για τα θέματα των διατλαντικών σχέσεων, της αμερικανικής παρουσίας στην Ευρώπη, τη συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία Τη συνεργασία που έχουμε στην καταπολέμηση της τριμοκρατίας, ε, τις προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας με τη Ρωσία και με τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Άρα το δικό μου έργο είναι πολύ πιο εύκολο και άρα μπορεί να είμαι πολύ πιο σύντομος, παραγωλο που θα θίξω εν συντομία ορισμένα από τα ζητήματα που αναδείξατε εσείς. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την άποψη του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία είναι βασικός εταίρος συνομιλητής σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να μιλήσω στα γαλλικά, αλλά κάποια στιγμή θα το γυρίσω και στα αγγλικά, γιατί έχω αγγλικές σημειώσεις. Επιτρέψτε μου καταρχάς να κάνω μια προκαταρκτική παρατήρηση, μια αρχική παρατήρηση, την οποία ε, δεν ανέφερε η Αλεξάνδρα με πολλές λεπτομέρειες, η οποία όμως μου φαίνεται πολύ σημαντική. Μιλώ για το μετασχηματισμό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας τα πέντε τελευταία χρόνια. Από την κρίση στην ε, τα μετασχηματίστηκε βαθύτατα το ΝΑΤΟ. Είχαμε την 70η επέτειο πριν από κάποιες εβδομάδες στο Λονδίνο, τη γιορτάσαμε και ε, σίγουρα τα 70 χρόνια ύπαρξης ε, της συμμαχία αυτής υπάρχει μια μόνιμη προσαρμογή και μεταμόρφωση του οργανισμού. Είχαμε το ψυχρό πόλεμο, τα Βαλκάνια, τη δεκαετία του 90 ε, είχαμε τα καθοριστικά στοιχεία και καθοριστικές χρονιές. Σήμερα η κατάσταση ε, την οποία βιώνουμε δεν είναι ίσως η πιο επικίνδυνη, αλλά ίσως είναι σίγουρα η πιο απρόοπτη καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ΝΑΤΟ, γιατί στην ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας βρίσκεται μια Ρωσία η οποία επιβεβαιώνει με όλο και περισσότερες δυνάμεις την στρατηγική ατζέντα που ακολουθεί, στρατηγική πολιτική ατζέντα. Έχουμε σε όλη την νότια πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ε, ε, μεγάλη αστάθεια και απειλές τρομοκρατίας και υβριδικές απειλές και κινδύνους. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο ε, για να μιλήσουμε για περίπλοκες απειλές. Και έχουμε και την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και την γρήγορη ανάδειξη στο προσκήνιο της Κίνας ως υπερδύναμης όχι μόνο στην Ασία αλλά ως μεγάλης δύναμης η οποία ε, προβλέπει να ε, καταλάβει όλο και μεγαλύτερο χώρο και στην ε, βόρειο-ατλαντική, αν θέλετε, επικράτεια. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τις απειλές και τους κινδύνους και προσαρμόζουμε αντιστοίχως τα αμυντικά μας εργαλεία και πρέπει όλα αυτά να τα ταιριάξουμε με το πιο σημαντικό με το να επαναπροσδιορίσουμε ε, και να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας για συλλογική άμυνα μέσα σε μία γενιά. Αυτή ήταν η αποστολή μας και έγινε ε, και έγινε πράξη μέσω διαφόρων πραγμάτων. Καταρχάς έχουμε εξυγχρονισμό των δομών διοίκησης και ελέγχου. Για πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου έχουμε ουσιαστική ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων διοίκησης και ελέγχου. Έχουμε ε, την ε, ενίσχυση της αντιδραστικότητας ε, των δυνάμεών μας, δηλαδή έχουμε δώσει έμφαση στη γρήγορη ανάπτυξη των δυνάμεών μας και έχουμε και ανάπτυξη των δυνάμεων στην Ανατολική ε, πτέρυγα της συμμαχίας των δυνάμεων που εδρεύουν στις χώρες της Βαλτικής και στην Πολωνία οι οποίες δυνάμεις, είναι σε οι οποίες δυνάμεις θα ήταν σε θέση, είναι πλέον σε θέση να δώσουν σημαντική ε, απάντηση μετά την κατάσταση στη Κρυμαία. Έχουμε και τις κυβερνοαπειλές και έχουμε και την ανάδειξη δυνάμεων στο διάστημα και ανακηρύχθηκε το διάστημα ως βασικός τομέας επιχειρησιακός για εμάς στο Συμβούλιο Υπουργών το Δεκέμβριο πέραν των, ε, ε, των, της θαλάσσιας οδού, της χερσαίας, της εναέριας οδού αλλά και της ε, διαδικτυακής επικράτειας και το διάστημα έρχεται να καθιερωθεί ως χώρο στον οποίο η Βορειοατλαντική Συμμαχία ε, θεωρεί ότι οφείλει να παρεμβαίνει. Αυξάνονται οι κυβερνοαπειλές περισσότερο από ποτέ. Είναι η μεγαλύτερη απειλή μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ο Γενικός Γραμματέας ε, αναφέρθηκε σε ένα νούμερο 130 εκατομμύρια δολάρια, 117 εκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα που ε, δαπανήθηκαν για την άμυνα από τους συμμάχους και τον Καναδά από το 2016. Είναι σημαντικό το ποσό. Ε, σε ετήσιο ρυθμό μιλούμε για μια αύξηση που μεταφράζεται με την ετήσια προσθήκη ε, ενός προϋπολογισμού ο οποίος θα ήταν αντίστοιχος με το ΑΕΠ μιας μεγάλης χώρας όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Άρα αυτά τα ποσά είναι σημαντικά οι προβλέψεις με βάση τα σχέδια που πρότειναν οι σύμμαχοι. Έχουν αθρηστική αύξηση της τάξης των 360 δις ευρώ που θα δαπανηθούν επιπρόσθετα από αυτά που δαπανήθηκαν την περασμένη δεκαετία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και έτσι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της απαξίωσης των ε, ε, εξοπλισμών μας. Δεν μιλούμε για μια κούρσα εξοπλιστική όπου θέλουμε να εξοπλιστούμε περισσότερο από τον άλλον. Μιλούμε για μια αντικατάσταση και επιδιόρθωση και ενημέρωση και επικαιροποίηση των εξοπλιστικών μας συμμάχων. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω στα αγγλικά και να πω το εξής. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αναλάβει μια δέσμευση εναντί στην Ευρώπη και αν θέλετε το συζητούμε αυτό και έχουν αυξημένο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και συχνά παραγνωρίζεται αυτό γιατί ξέρετε τίνουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην πολιτική ε, συζήτηση που γίνεται για το μοίρασμα των βαρών. Όμως οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν περισσότερα στρατεύματα και κάνουν περισσότερη εκπαίδευση και είναι πιο παρούσες στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα σήμερα παρά τα παλαιότερα χρόνια. Φέτος έχουμε τον Defender 24. Είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ε, έγινε σύνοδος υπουργών στα, στις αρχές Δεκεμβρίου με πολύ αίσια έκβαση. Ήταν σαφές ότι οι, οι συζητήσεις μεταξύ συμμάχων παραμένουν έντονες και εσείς κυρία Πρόεδρε και η Αλεξάνδρα αναφέρθηκατε σε αυτό. Οι συζητήσεις στρέφονται γύρω από τρία ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να θίξω εν συντομία. Το μοίρασμα των βαρών, ο στόχος του 2%, burden sharing, να αντιστοιχεί στο βαθμό της προσπάθειας ε, στο μέσο όρος του ψυχρού πολέμου ήταν 3%. Δεύτερον, συζήτηση ε, για το κατά πόσο που βρίσκονται ε, για το κατά πού βρίσκονται οι μεγαλύτερε απειλέ και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μα αντίπαλοι. Υπήρχαν κάποιε διαφορέ απόψεων, αλλά είναι παραπλανητικό να θεωρούμε ότι υπάρχει διαίρεση μεταξύ αυτών που νομίζουν ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι στα ανατολικά και οι άλλοι που νομίζουν ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι στα νότια. Δεν ισχύει αυτή η διαίρεση γιατί και η Ρωσία είναι εξαιρετικά δραστήρια στα νότια, ενώ η τρομοκρατία για παράδειγμα δεν γνωρίζει σύνορα και αυτό το έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένω. Τώρα, Πώς θα ενισχύσουμε τη συνοχή μεταξύ των συμμάχων. Δεν έχει τελειώσει η προσαρμογή και ο μετασχηματισμός του ΝΑΤΟ, της Φοροατλαντικής Συμμαχίας. Θα συνεχίζουμε αυτά Είναι μια διαδικασία προβληματισμού περί συλλογής, την οποία ξεκινήσαμε στο Λονδίνο, την οποία θα οριστικοποιήσουμε τους επόμενους μήνες. Η Συμμαχία εξετάζει τους βασικούς πολιτικούς κανόνες ε, και πώς μπορούν να ενισχυθούν, ε, να ενισχυθούν οι δεσμοί με βάση αυτούς. Η προσαρμογή αυτή δεν λαμβάνει χώρα εν κενό. Και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Παρά που εμείς ε, έχουμε την έδρα μας στο ΕΒΕΧ στις Βρυξέλλες, το ΝΑΤΟ εκεί έχει την έδρα του σε αυτή τη συνοικία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε στο χρυσελεφάντινο πύργο μας και ότι ε, λειτουργούμε εν κενό τελείως αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει την έδρα της εδώ στο Έτερμπεκ. Ε, συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Έθνη και με τους λοιπούς, με τις σκανδιναβικές χώρες. Και όπως σας είπε και ο Γενικός Γραμματέας την Τρίτη, έχετε δει και τις δύο πλευρές του ίδιου ε, νομίσματος. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια ε, συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ με ε, κοινέ δηλώσεις που έχουν υπογραφεί από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γιούνκερ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Τούσκ με την προηγούμενη σας με την προηγούμενη Επιτροπή. Η συνεργασία αυτή δεν είναι πάντοτε εύκολη. Όμως, τρία χρόνια είμαι σε αυτή τη θέση και έχω δει τεράστια πρόοδο να σημειώνεται προς αυτή την κατεύθυνση κάθε εβδομάδα. Έχω συνεργασία με Ευρωπαίους ομολόγους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, είτε πρόκειται για στρατιωτικά θέματα, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διάφορες γενικές διευθύνσεις της. Όλο και περισσότερο έχουμε συνεργασία καθημερινή και εβδομαδιαία. Τώρα, Πώς οι τρίτες χώρες αλληλεπιδρούν με τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια ζητήματα μπορεί να είναι λεπτά για συμμάχους που είναι μέλη του ΝΑΤΟ αλλά δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι με καλή βούληση λύνονται τα ζητήματα και μάλιστα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Όμως αυτή αυτό το θέμα θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία τα, τα επόμενα χρόνια και πρέπει να δουλέψουμε πάνω στις ικανότητες, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές. Η συζήτηση για την Κίνα, στην οποία αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα, αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το περιβάλλον του ΝΑΤΟ είναι το πλέον κατάλληλο για να ε, λυθεί το θέμα αυτό. Όταν γίνεται λόγος για την πέμπτη γενιά, τα δίκτυα πέμπτης γενιάς και για το quantum computing, 5G and quantum, ε, quantum computing, κβαντική υπολογιστική. Ε, πρέπει να είμαστε σε θέση να τα συζητούμε αυτά και να είμαστε προετοιμασμένοι σε ένα ταχαίως εξελιζόμενο, σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Εμεί ε, στο ΝΑΤΟ αντιπροσωπεύουμε το μεγαλύτερο μέρο τη παγκόσμιας οικονομία και το μεγαλύτερο μέρο τη ε, παγκόσμιας ε, στρατιωτικής ισχύω. μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προς το συμφέρον όλων να συνεργαζόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις μαζί, από κοινού. Για να ολοκληρώσω, εν συντομία, να πω το εξή. Για να έχουμε ισχυρή άμυνα, πρέπει να συνεχίσουμε να εξυγχρονίζουμε το, τα μέσα μας και να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ΝΑΤΟ εμείς πιστεύουμε, είμαστε υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας και περιμένουμε πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει πιο δραστήρια σε αυτό το τομέα. Αν το κάνει σωστά θα υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις στην άμυνα, θα υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες ε, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνει πιο δίκαιο μοίρασμα και τελικά θα καταστεί ισχυρότερη η συμμαχία. Άρα πρέπει να ταιριάξουμε το υψηλό επίπεδο της στρατηγικής ε, συνεργασίας με το υψηλό επίπεδο των φιλοδοξιών που έχουμε όλοι θέσει και αυτό να φανεί και στη πράξη. Να μοχλεύσουμε λοιπόν αυτά τα εργαλεία για να αποκομίσουμε τη μέγιστη ε, προστιθέμενη αξία, πάντοτε διατηρώντας ρεαλισμό, κοινή λογική, κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο όπως γνωρίζετε και κάτι το οποίο όμως πρέπει να δουλεύουμε ε, καθημερινά. Με αυτά και με αυτά, επιτρέψτε μου να ε, ολοκληρώσω την παρέμβασή μου κάπου εδώ, ευχαριστώντας για άλλη μια φορά εσάς κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, για την πολύ ευγενική σας πρόσκληση. Παραμένω στη διάθεση των παριστάμενων για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση και για να τοποθετηθώ και πιο συγκεκριμένα για θέματα του χαρτοφυλακίου μου των αμυντικών επενδύσεων. Στόχος μου είναι να προωθήσω την συνεργασία με ε, έμφαση στην τεχνολογία και την πυραυλική άμυνα. Θα ήταν ένα παράδειγμα απλά που σας ε, δίδω, ε, εάν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Η Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο στους διαφόρους συναδέλφους, θα ήθελα να σας προτείνω να μην ολοκληρώσουμε στις 12, αλλά να καθίσουμε λίγο παραπάνω για να μπορεί να υπάρξει αληθινή ανταλλαγή απόψεων και ερωτήσεις και απαντήσεις. Όσοι μπορείτε να καθίσετε και μετά τις 12 αν ε, μπορείτε να καθίσετε γιατί έχουμε τους δερμηνείς μέχρι τις 12.30. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε λοιπόν ε, αυτό το χρονικό διάστημα. Ο κύριος Κρίς Πίτερς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω την ε, κυρία Χοψεφέρ και τον κύριο Γκρόν για, για τα όσα μας είπαν σήμερα σε αυτήν την συνεδρίαση τον Απρίλιο. Ε, θα έχουμε την επέτειο των 70 χρόνων του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρί, υπογραμμίσουμε την σημασία της ε, συμμαχίας ευελπιστώντας ότι η συμμαχία θα ισχύει ακόμα ε, και σε 50 και σε 100 χρόνια από σήμερα. Ε, βεβαίως αξιολογούμε πολύ θετικά την ε, συμμαχία. Η συμμαχία και το ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το σλόγγαν της συμμαχίας είναι «Atmos in consulento liber» στα λατινικά, στα γαλλικά πώς να το πω. Ε, το πνεύμα είναι ελεύθερο, ε, ενδιαβουλεύσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ε, σαν αρχή σε αυτούς τους καιρούς που καλούμαστε να βρούμε αποφάσεις, συγγνώμη, απαντήσεις στα νέα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, να σας ε, υποβάλω όσον αφορά ε, την συμμετοχή στο, στη συμμαχία. Δηλαδή τα νέα μέλη Υπάρχει εδώ ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο προκύπτει. Ε, άλλωστε πριν από λίγο καιρό πήγαμε στο Κίεβο στην Ουκρανία. Η ερώτησή μου είναι ποια είναι πλέον αυτή τη στιγμή η θέση του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ουκρανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από ό,τι κατάλαβα, το 2008 ε, είχε πει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα ανοίξω το ΝΑΤΟ και προς την Ουκρανία και ήταν ε, ε, πολύ θετική η ανταπόκριση. Όμως τώρα είμαστε σε διαφορετικές ε, καταστάσεις. Έχουμε και το πρόβλημα του ε, Ντόνες και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε ποια είναι η νέα θέση. Αναφερθήκατε άλλωστε ε, κύρια μου και στο θέμα της ε, Μέσης Ανατολής. Βεβαίως εδώ δεν προκύπτουν ζητήματα μέλους, ελπίζω, αλλά δεν αποκλείεται τίποτα. Δεύτερον, τι θα κάνουμε με τα, ας τα ονομάσουμε δύσκολα μέλη. Και εδώ η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, προκύπτει το ζήτημα και με, το, με την Τουρκία. Ξέρω το, για το ΝΑΤΟ είναι σημαντικό μέλος η Τουρκία, αλλά έχω πολλούς συναδέλφους που είναι πεπισμένοι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο μέλος της συμμαχίας η Τουρκία. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με αυτό το ζήτημα της Τουρκίας, ποιος θα είναι ο μελλοντικός ρόλος της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ κλπ. Τρίτη ερώτηση ε, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα την ευκαιρία να υποβάλλω το ερώτημα αυτό στο Γενικό Γραμματέα η αντιπροσωπεία με το ΝΑΤΟ είναι πολύ συγκεκριμένη αντιπροσωπεία. Βεβαίως εμείς έχουμε και πολλές ε, φιλοδοξίες, άλλωστε έχουμε και καινούργια στοιχεία, έχουμε το EDF και νομίζω ότι ήρθε η ώρα ε, να αναβαθμιστεί η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τελειώνοντας, δεν θα έχουμε άνιμους συνκονσουλέν του Λίμπε, αλλά άνιμους Ευρωπαία, ευρωπαϊκό πνεύμα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τον λόγο ε, στον ε, Σβέν Μίξερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για τις πλήρες παρουσιάσεις σας, ενδελεχείς παρουσιάσεις σας. Δεν έχω ερωτήσει ακριβώς, σχόλια περισσότερο έχω να κάνω. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι η αντίληψη της συλλειτουργίας ε, του ΝΑΤΟ διαφέρει αν το βλέπει κανείς από την ε, πλευρά των ΗΠΑ ή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, βεβαίως, ναι, είναι γεγονός ε, ότι από την πλευρά των ε, ε, Ηνωμένων Πολιτειών υπήρχε πάντα αυτή η αντίληψη της ασφάλειας από τον ψυχρό πόλεμο και μετά. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει μία αποτελμάτωση πνευματική και επιχειρησιακή η, η εδαφική ας πούμε ακαιρεότητα ή η άμυνα, η εδαφική το, τον του ευρωπαϊκού εδάφους έχει ολοκληρωθεί κατά κάποιο τρόπο ως αποστολή ε, ε, ε, και υπάρχει πλέον μία αποτελμάτωση. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν Εγώ 20 χρόνια ασχολήθηκα, 15-20 χρόνια με την εθνική πολιτική και ήμουν ε, και για 15 χρόνια μέλος ε, της ε, ε, ε της Συνέλευσης και βεβαίως εκεί χρησιμοποιούσαμε, μιλούσαμε ε, σύρι, κυρίως για χερσαίες δυνάμεις, εκ των οποίων το 5 8% ήταν άμεσα διαθέσιμο ε, για ε, να ε, χρησιμοποιηθεί επιτόπου μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Έκτοτε, Βεβαίως έχουμε μειώσει την φιλοδοξία όσον αφορά αυτού του είδους της εμπλοκές. και επομένως δεν υπάρχει πραγματικά δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης. Ε, εμείς ε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα λέγαμε ότι είμαστε έτοιμοι ε, για οποιασδήποτε εμπλοκές. Τώρα μιλάμε περισσότερο για transformation exercises. Βεβαίως, όταν αναφερόμαστε σε παρουσία αμερικανικών δυνάμεων σε ευρωπαϊκό έδαφος, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερες δυνάμεις. Επίσης γίνονται κοινέ ε, επιχειρήσεις ή κοινέ ασκήσεις περισσότερο με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ωστόσο υπάρχει πάντα σκεπτικισμός των Ευρωπαίων σχετικά με την εμπλοκή των Αμερικανών στην Ευρώπη. Και γενικώ ε, υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον μπορούμε να βασιστούμε στους Αμερικανούς και ότι αυτοί θα κάνουν το σωστό γιατί αναλαμβάνονται και βήματα τα οποία εκφεύγουν της ε, πολιτικής άμυνας. Δεν το ξέρω ότι δεν είναι πραγματικά ερώτηση, αλλά ωστόσο είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να λησμονούμε και να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και σε μελλοντικές αναλύσεις της συνεργασίας. Merci. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπασέσκου. Well, Ευχαριστώ πολύ ε, για τις εξαιρετικές ε, παρουσιάσεις ε, που μας κάνατε. Έχω και εγώ μερικά σχόλια. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι εντός του ΝΑΤΟ υπάρχει μια κρίση έλλειψης κατανόησης. Δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι πιο γρήγορη η Ευρωπαϊκή Ένωση ή, ε, ή, ή το ΝΑΤΟ όσον αφορά τις, ε, τα νέα μέλη. Αναφέρομαι και στην Βόρεια Μακεδονία εδώ. Είχαμε από το 2008, όπως είπε και ο συνάδελφος που ξεκίνησε η ιστορία της ε, Ουκρανίας. Γινόταν λόγος για, για την Ουκρανία και την Γεωργία που πήραν τον οδικό χάρτη για την προσχώρηση, για την ένταξη. Μετά είχαμε αντιδράσεις ε, από άλλες ε, ε, χώρες και περιοχές και από την Γερμανία που προσπαθήσαμε επί ώρες να πείσουμε την Άγγελα να πει ναι, αλλά παρόλα αυτά εισπράξαμε ένα βροντερό όχι. Επομένως, εξακολουθεί η ίδια ιστορία πήρανε τον οδικό χάρτη στο Βουκουρέστι, αλλά χάθηκε μια ευκαιρία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει έλλειψη κατανόησης. Ε, Από την ευρωπαϊκή πλευρά, η Ευρώπη λέει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν μειώσει την παρουσία τους στην Ευρώπη. Φυσικά, αφού πρέπει να καλύψουν τις εξελίξεις από την Ασία και στον Ασία και τον Ειρηνικό. Εν μία νυχτή ανακάλυψαν ότι η Βόρεια Κορέα είναι πυρηνική, έχει πυρηνικό ε, οπλισμό και ε, ότι η Κίνα πλέον είναι διαφορετικός πέκτης και από τη στιγμή που είδαν ε, στην Κίνα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ρωσία βρίσκονται πλέον ας πούμε στην ίδια γραμμή άρχισαν να αναπτύσσουν το πλωστάσιό τους. Η ερώτηση μου λοιπόν και μη με θεωρήσετε φιλοαμερικανό παρακαλώ εγώ απλώς προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Εμείς λέμε ότι έφυγαν οι Αμερικάνοι, μείωσαν την παρουσία τους στην Ευρώπη, ενώ από την άλλη πλευρά δεν ξέρω καμία ευρωπαϊκή χώρα η οποία να υποστηρίζει την Αμερική στις δραστηριότητές τους στην Ασία και τον Ειρηνικό. Δεν έχει πολύ λογική αυτό. Δεν έχω δει καμία χώρα ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίζει ε, την, ε, συνωμένες Πολιτείες, ε, στην Ασία και τον Ειρηνικό. Επίσης, ε, στην διάσκεψη του 14 στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπαμε, καθορίσαμε ότι το ΝΑΤΟ ε, θα δώσει εξοπλισμό ε, στα νότια ανατολικά ε, σύνορα του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Έγινε αυτό. Είναι πολύ ενεργή στα ανατολικά σύνορα. Δεν βλέπω όμως πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της Ευρώπης. Βλέπω όμως πολλές αμερικανικές βάσεις οι οποίες ξεφυτρώνουν κάθε χρόνο. Στη Ρουμανία να σας πω έχουν τώρα ξεκινήσει την τρίτη αεροπορική βάση ε, η οποία ανήκει ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κοινέ ασκήσεις, τουλάχιστον μία το χρόνο στην Ανατολική Ευρώπη και στα Ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι εν τέλει, όταν λέμε θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, έρχονται. Θυμάμαι όταν η Washington αποφάσισε να μειώσει την παρουσία της στην ε, κεντρική Ασία έτσι ώστε να καλύψει ε, την Ασία ειρηνικό, αλλά δεν έχουμε την ειλικρίνεια να παραδεχτούμε ότι θα κάνουμε την προσπάθεια να συμβάλλουμε με 2% ε, στους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Εδώ ο Τραμπ είναι businessman, είναι έμπορος και επομένως δεν εφαρμόζει καθαρά πολιτική σε αυτό το θέμα. Σκέφτεται δηλαδή όχι σαν πολιτικός αλλά σαν businessman. Εμείς έχουμε συμβολή 1,41% του ΑΕΠ, δηλαδή ε, μείον 90 δις το χρόνο. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο. Από τη μία μεριά να ζητάμε από τις Ευρω... Πολιτείε Πολιτείες να μας ε, προστατεύουν και να δίνουν το 3,3% του ΑΕΠ και να καθιστούν προτεραιότητα, ας πούμε, ε, το δικό μας βιωτικό επίπεδο εδώ στην Ευρώπη. Δηλαδή να λέμε στους Αμερικάνους ελάτε να μας ε, ε, προστατέψετε γιατί εμείς δεν θέλουμε να δίνουμε αυτή τη συμβολή να συνεισφέρουμε το 2%. Εδώ υπάρχουν προβλήματα κατανόησης λοιπόν. Πέραν αυτών δεν θεωρώ παρόλα αυτά ότι έχουμε κάποια καλύτερη λύση για την άμυνα και για την ασφάλειά μας. και την, πώς να σας το πω, Δεν συμφωνώ με αυτόν τον όρο, στρατηγική αυτονομία. Πώς μπορεί κανείς να είναι αυτόνομος στρατηγικά, όταν δεν έχεις τη δυνατότητα, όπως δεν έχει η Ευρώπη, να διατηρήσεις ε, την παγκόσμια ισορροπία. Αυτό γίνεται μονάχα από την Κίνα, τη Ρωσία και τις Ηνωμένε Πολιτείε, από αυτές τις τρεις χώρες. Και δεν είναι δυνατόν εδώ τώρα να συζητούμε για οικονομικές δυνάμεις, γιατί η Ρωσία δεν είναι οικονομική δύναμη. Έχει μικρότερο ΑΕΠ από την Ιταλία. Ωστόσο είναι global player διότι έχουν πυρηνικό οπλοστάσιο. Αγαπητέ συνάδελφε, λέει η πρόεδρος, ε, ε, είναι και άλλοι που θέλουν να πάρουν τον λόγο. Εκ μέρου του ID, ο κύριο Μάντισον, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τα πολλά και ενδιαφέροντα. Ε, εν πολύ συμφωνώ με αυτά που είπατε. Συμφωνώ και με τον προηγούμενο μιλητή, με τον αγαπητό συνάδελφο από τη Ρουμανία. Μου λέτε ότι δεν υπάρχει καλύτερο αμυντικό σύστημα από αυτό που έχουμε σήμερα, το ΝΑΤΟ δηλαδή. Έχω κάποια ερωτήματα. Η κυρία από το Marshall Fund από το Παρίσι είπε αρκετέ φορέ ε, ότι κινούμεθα σε μια νέα παγκόσμια κατάσταση. Όντως και υπάρχει πολυφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε αυτονομία. Υπάρχουν όμως νέοι κίνδυνοι που προκύπτουν από την Κίνα, Ρωσία, Μέση Ανατολή. Και είναι ξεκάθαρο ότι η αυτονομία από τη ΣΥΠΑ σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε, χωριζόμαστε. Δηλαδή σαν μια μεγάλη δύναμη αποχωριζόμαστε. Γιατί μιλάμε συνεχώς για αυτονομία. Υπάρχει κάποιος πολιτικός λόγος. Αν το δούμε σήμερα, τρία χρόνια μετά την νίκη του Τραμπ στις εκλογές, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη. Πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Πολωνίας και ΕΠΑ, Εστονίας και ΕΕ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ για θέματα άμυνας. Σε μερικές περιπτώσεις Μπορεί να ήταν και έξυπνη κίνηση του Τραμπ που έθιξε το θέμα των δαπανών, γιατί τώρα πολλές χώρες το σκέφτονται και μας τρομάζει λίγο. Οι δράσει των ΗΠΑ στο Ιράκ και στο Ιράν ε, δεν έχουν τίποτα καινούριο και το 2003 στο Ιράκ το είδαμε και με άλλες κυβερνήσεις των ΗΠΑ. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντοτε 100%, αλλά το θέμα είναι τι είναι καλύτερο, τι είναι χειρότερο. Τώρα νομίζω ότι είναι καλύτερα να υποστηρίζουμε τους συμμάχους μας όταν καταπολεμούμε την τρομοκρατία και τη ρίζοσπαστικοποίηση ε, και την μεγάλη άσκηση επιρροής από άλλες χώρες. Δεν ξέρω γιατί συζητάμε λοιπόν τόσο πολύ το θέμα της αυτονομίας και των διαφορών μας με τους Αμερικανούς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η αλληλεγγύη μέσα στο ΝΑΤΟ. Αλλά πώς βλέπουμε τα πολιτικά προβλήματα από της Γαλλία και Γερμανίας. Αν ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν, ε, είπε, όπως είπε αρχές Δεκεμβρίου ότι χρειαζόμαστε μια νέα έναρξη των οικονομικών σχέσεων με την ε, Ρωσία. Ε, αυτό τι σημαίνει, μήπως έχουμε στο οπτικό μας πεδίο την Ουκρανία και αλλάζει κάπως η κατάσταση σε σχέση με τη Ρωσία. Επίσης είπε ο κ. Μακρό ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό το ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό για τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ και για τα οικονομικά συμφέροντα μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, αν δούμε το Nord Stream 2, που μπαίνουν. Γιατί όταν μιλάμε για αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε την ίδια κατανόηση της ε, άμυνας και των κοινών μας συμφερόντων. Αν το βλέπουμε όμως διαφορετικά και αν οι Γερμανοί δεν ενδιαφέρονται για τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των συμμάχων τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θέλουμε να αγοράσουμε φθηνό αέριο από τη Ρωσία και δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλες χώρες που φοβούνται λίγο αυτή την επιρροή στην ενεργειακή πολιτική. Αυτό τι σημαίνει για την αυτονομία και τη συνεργασία και στα αμυντικά συστήματα. Οι δύο μιλητές νομίζω ότι το βλέπουν διαφορετικά γιατί ο κύριος Γκραντ είναι από το ΝΑΤΟ, η κυρία προέρχεται από το Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ, αλλά θα ήθελα να έχουμε μια εικόνα. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, λέει η Πρόεδρος, ο κ. Σατόρη πολύ γρήγορα. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η απάντηση του ΝΑΤΟ για την διάδοση των όπλων και των πυρηνικών πυράβλων. Έχει διαμορφωθεί κάποια απάντηση. Ποια είναι η στρατηγική στο θέμα αυτό. Δεύτερον, η στρατηγική αυτονομία μου φαίνεται εξαιρετική έννοια. Αλλά πώς ε, εντάσσεται σε όλα τα στάδια των σχέσεών μας με τη ΣΥΠΑ. Με τον Τραμπ βλέπουμε ένα παροξισμό των ΗΠΑ. Βλέπουμε μια υπαναχώρηση σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Πώς θα επανέλθουμε σε ισορροπία μέσα στο ΝΑΤΟ με μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση με στρατηγική αυτονομία που θα εντάσσεται όμως στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ. Δεν μιλάμε μόνο για τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ στον κόσμο, αλλά χρειάζεται και μια επανισορροπία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Και αυτό πώς το αναλαμβάνουμε από οικονομικής πλευράς. Και αν θέλουμε να έχουμε αυτονομία της Ευρώπης, τη δεύτερη πτυχή που περιγράψατε, πώς θα το κάνουμε. Πολύ συγκεκριμένα στην πράξη με στρατιωτική συνεργασία ισχυρότερη μεταξύ Ευρωπαίων και στην πράξη πώς διαρθρώνεται. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό στρατό και τι μορφή θα έχει. Όπως ο στρατός του ΝΑΤΟ ε, υπάρχει στην πράξη μέσα στο ΝΑΤΟ. Και τελικά μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ενότητα, στρατηγική ενότητα, διπλωματική ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά δεν βλέπω πώς εντάσσονται μέσα στις σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ. Επίσης, στις σχέσεις μας και με άλλες, μεγάλες, και με άλλες δυνάμεις, ε, επί ποιες βάσεις θα γίνει αυτό. Υπάρχει ε, η πολιτική εικόνα, υπάρχουν οι ευρωπαϊκές αξίες, γιατί υπάρχουμε και εκτός ΝΑΤΟ και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και σε σχέσεις με άλλους και δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τις αξίες μας. Και ως οικολόγος βλέπω ότι έχουμε απέναντί μας ένα Αμερικανό πρόοδο που αρνείται την ύπαρξη κλιματικής αλλαγής. Αυτή την αποσταθεροποίηση πώς θα την εκλάβουμε σε σχέση με τις πολιτικές μας επιλογές και με τις αξίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον Καμί καταρχήν και μετά στην Αλεξάνδρα Ντεχόφουσέφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που μας στέθηκαν. Θα είμαι αρκετά λακωνικός και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όσον αφορά τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, η συμμαχία έχει επεκταθεί και συνεχίζει να επεκτείνεται. Σύντομα θα έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία που είναι σημαντικό βήμα. Το Μαυροβούνιο εντάχθηκε το 2017. Έχουμε μια πολιτική ανοιχτών θυρών που δουλεύει στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Για την Ουκρανία και τη Γεωργία παραμένουν ανοιχτά τα θέματα. Υπάρχει το σχέδιο δράσης όπως αποκαλείται βάσει του οποίου καταβάλλεται μια προσπάθεια να προσφέρουμε στις χώρες αυτές μια πιο στενή σχέση με τη συμμαχία που να λειτουργεί και στην πράξη. Ήμουν επικεφαλής ε, της ομάδας τεχνικής συνεργασίας με τους Ουκρανούς Έχουμε συχνά συνεδριάσεις ε, και κάνουμε πολλά σε σχέση με τους Ουκρανούς. Δηλαδή γίνονται πολλά πράγματα για να έχουμε μια πιο στενή εταιρική σχέση. Όσον αφορά το αν θα γίνουν μέλη, αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η Συμμαχία εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Και πάντοτε γίνεται μια συζήτηση στη Συμμαχία όταν τίθενται θέματα για νέα μέλη, ιδίως όταν πρόκειται για χώρες για τις οποίες υπάρχει και κάποια ε, σύγκρουση. Το Βορειοκρατικό Σύμφωνο επισκέφθηκε και τη Γεωργία και την Ουκρανία πέρυσι και γίνονται συνεχώς ανταλλαγές απόψεων ε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΝΑΤΟ Ουκρανίας και της Επιτροπής ΝΑΤΟ Γεωργίας. Συνεχίζονται λοιπόν οι συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Η έννοια της εταιρικής σχέσης αφορά ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα γειτονικά κράτη, αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής. Η παρουσία μας στο Κουβέιτ είναι μια ευκαιρία να έχουμε συνεργασία με τις χώρες του κόλπου, έχουμε στενή συνεργασία με την Ιορδανία, με πολλές ευκαιρίες στη συνεργασία μας. Πολλά γίνονται λοιπόν και σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θέλω να αναφερθώ σε κανένα σύμμαχο ως δύσκολο σύμμαχο, αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιες χώρες στη συμμαχία που ε, υπεραμείνονται των θέσεών τους με μεγάλη ένταση. Η Συμμαχία λειτουργεί με τον κανόνα της συνένεσης και επιμένουμε σε αυτό. Θέλω να σας πω ξεκαθαρά ότι στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο γίνονται πολύ έντονες συζητήσεις και πολλές χώρες έχουν ε, ισχυρές εθνικές θέσεις τις οποίες υπερασπίζονται ή έρχονται και επικρίνουν άλλους συμμάχους για τις πράξεις τους στο ε, Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Και για τα γεγονότα στη Συρία, παραδείγματο χάρη, έγιναν πολύ ανοιχτέ και έντονε συζητήσεις στι συνεδριάσει του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Κάτι που θα συνεχιστεί. Όλοι οι σύμμαχοι συμμετέχουν. Κάποιοι ακούγονται ε, περισσότερο, κάποιον οι φωνές ακούγονται περισσότερο ε, και για το θέμα της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος και γεωγραφικά καταρχήν και λόγω μεγέθους και είναι ένας σύμμαχος που πάντοτε πολύ ξεκάθαρα υπεραμείνεται των θέσεων τους στη συμμαχία. Για την κοινοβουλευτική διάσταση, εγώ ε, προσπαθώ να συνεργάζομαι συχνά με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι πάντοτε έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούν και ενδιαφέρονται. Και όταν μιλάμε για δαπάνε, πρέπει να συζητούμε είτε με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, για να μπορέσουμε να κάνουμε αποδεκτά αυτά τα οποία προτείνουμε. Είναι μια πολύ σημαντική διάσταση, λοιπόν, η διακοινοβουλευτική συνέλευση. Επομένω, είναι σημαντικό εταίρο. Ο πρώτο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έλεγε ότι προσπαθούσαν να κρατήσουν μέσα τους Αμερικανούς, έξω τους ε, Ρώσους ε, και ε, να κρατήσουν πιο χαμηλά τους Γερμανούς. Δεν ξέρω τώρα ποιος προσπαθεί να δαπανά περισσότερο. Έχουν εξελιχθεί οι απόψεις με το πέρασμα του χρόνου, δαπάνες για διάφορες παρεμβάσεις. Κάτι που ανέφερε η Αλεξάνδρα είναι η έννοια της στρατηγικής παράλυσης. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση και γίνονται πολλά για το θέμα αυτό και προσπαθούμε να συμβαδίζουμε με τα γεγονότα που συμβαίνουν παγκοσμίω. Μερικές φορές τα καταφέρνουμε καλύτερα, μερικές φορές είναι πιο δύσκολο. Τελικά όμως αυτό είναι ο στόχος της συμμαχίας. από αυτά που είπατε για την ετοιμότητα και για τη χρησιμότητα όλων των δυνάμεων. Θα ήθελα να πω ότι επικεντρωνόμαστε στο ρόλο της αλλαγής. και για το σεισμό στο Πακιστάν ε, βοηθάμε με δυνάμεις ε, του ΝΑΤΟ και υπάρχει έμφαση για τη διαλειτουργικότητα, για το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε μαζί επιχειρησιακά και να έχουμε κοινή εκπαίδευση. Η ετοιμότητα συμφωνήθηκε και από τους συμμάχους πέρυσι. Έχουμε 30 τάγματα και 30 σκάφη διαθέσιμα σε 30 μέρες ή λιγότερο. Ε, και αυτό είναι μια έννοια που έχει άμεση σχέση με την πραγματική μας επιχειρησιακή δυνατότητα, να μην ε, παραμένουμε σε δεσμεύσεις, αλλά να έχουμε κάτι το οποίο μπορεί στην πράξη να εκδιπλωθεί πολύ γρήγορα. Για την παρουσία των ΗΠΑ, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως έχει εξελιχθεί κατά πολύ η παρουσία των ΗΠΑ. Δεν υπάρχουν τα στρατεύματα που υπήρχαν την εποχή του ψυχρού πολέμου στην Ευρώπη. Τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα και από την άλλη πλευρά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε και η παρουσία σε μερικές περιπτώσεις ε, είναι σημαντική για να προχωρούμε η εντύπωσή μου είναι ότι έχει αυξηθεί η παρουσία των ήπα και δεν είναι απλώς εντύπωσή μου, είναι και πραγματικότητα. Επαναξιολογούμε τις προτεραιότητες και εξελίσσονται τα πράγματα. Όσον αφορά ε, τις χώρες ε, Ασίας και Ειρηνικού και την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουν οι Ευρωπαίοι. Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν ε, μια επιχείρηση ελεύθερης ναυσιπλοείας στη νότια θάλασσα της Αυστραλίας. Ίσως είναι μια δράση που πρέπει να επεκταθεί γιατί και αυτό είναι μια μορφή κατανομής βαρών σε τομείς όπου ηγούνται, σε περιοχές όπου ηγούνται οι Ηνωμένε Πολιτείε. Σχετικά με το ερώτημα για το 2%, αλλάζουν και πάλι τα πράγματα. Είχαν αναλάβει τη δέσμευση τρει εταίροι, τώρα είμαστε 7 και σύντομα 8. και έχουν αναλάβει τη δέσμευση μέχρι το 2024 ώστε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που αναφέραμε. Έχει αλλάξει δηλαδή και το ύφος της συζήτησης για το θέμα αυτό. Μπορεί να μην δεσμεύονται για 15% αλλά μπορεί να έχουν αναλάβει άλλες δεσμεύσεις σε άλλα θέματα κάποια εταίροι. Για τις διατλαντικές σχέσεις τώρα. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για τις διατλαντικές σχέσεις και στο παρελθόν. Δεν ξεκίνησε με τη συνέντευξη στο Economist, αλλά αυτές οι συζητήσεις γίνονται από πάντοτε, γιατί όλες οι χώρες είναι δημοκρατικές χώρες και οι ηγέτες έχουν ισχυρές προσωπικότητες και απόψεις. Από τη διάσκεψη του Λονδίνου μπορώ να πω ότι κατέληξε σε μια κοινή συνεννόηση για το τι πρέπει να γίνει μεταξύ άλλων ε, και σημαντική όθηση για διάλογο σε πολιτικά ζητήματα. Δεν υπάρχει έλλειψη ενότητας, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου. Παρότι και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, όταν συζητάμε το τι πρέπει να κάνουμε στη Μέση Ανατολή, τι κάνουμε με την πρόκληση της Ρωσίας, είναι φυσιολογικό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις ε, με βάση και την ε, γεωγραφική θέση των χωρών. Τελικά όμως, τα σχόλια τα οποία ε, προκύπτουν και οι συνεντεύξεις δεν εμποδίζουν το να έχουμε κοινή κατανόηση για τις στρατηγικές προκλήσεις και για τον τρόπο αντιμετώπισης τους από τη Συμμαχία συνολικά με όλους τους εταίρους συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις ε, όσο πιο σύντομα μπορούσα. <laughs> Τώρα εσεί έχετε το λόγο πιο ελεύθερα, γιατί μάλλον έχουν όλα υποθεί. Πράγματι, δύο δευτερόλεπτα θέλω να σταθώ σε αυτή την πολύ ε, ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να σταθώ δηλαδή στο θέμα της στρατηγικής αυτονομίας και τον αμερικανικό παράγοντο. Σύμφωνο με τον Καμίγ, δεν είμαστε ε, στη φάση της αμερικανικής απόσυρσης, αλλά σε μια εκ νέου εξισορρόπηση, εκ νέου ανάπτυξη των στρατιωτικών του δυνάμεων στο παγκόσμιο στερεώμα για να ε, επικεντρωθούν σε αυτό που θεωρούν πιο σημαντικό που είναι ο ανταγωνισμός με την Κίνα και αυτό θα έχει επιπτώσεις για εμάς τους Ευρωπαίους γιατί ε, αναπτύσσουν εκ νέου την παρουσία τους στην νότια πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, δηλαδή στην Αφρική και στην Ανατολή. Και η Ευρώπη αναπροσδιορίζει την δέσμευσή της στο Σαχέλ, ακριβώς γιατί θέλει να ε, ακριβώς εν ώψη της μερικής απόσυρσης των Αμερικανικών στρατευμάτων με σκοπό να στηρίξει την καλική αποστολή στο Σαχέλ. Δεύτερο θέμα είναι το εξής. Με δυσκολεύει η εξής ιδέα ότι δηλαδή η η στρατηγική αυτονομία σημαίνει απόσχηση και ανεξαρτητοποίηση από τους Αμερικανούς ή από την Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν είναι επί τούτου, δεν είναι περί αυτού. Ε, εάν πραγματικά θεωρούμε ότι πρέπει να αποσχιστούμε για τους Αμερικανούς, γιατί θεωρούμε ότι όντως δεν μοιράζονται τις αξίες μας ή δεν μοιράζονται την ίδια αντίληψη και ερμηνεία που έχουμε για την κατάσταση και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει έτσι να λειτουργούμε. Να έχουμε στρατηγική αυτονομία γιατί θέλουμε να κάνουμε τι, γιατί θέλουμε να έχουμε πια εργαλεία και μέσα για να πετύχουμε τι. Σε αυτό το ρώτημα πρέπει να απαντήσουμε. Έχουμε προσπαθήσει να παρεύουμε στη Συρία, στη Λιβύη, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί με Αύριο οι Αμερικανοί θα μας πούνε ότι κοιτάξτε για τη Συρία και τη Λιβύη δεν είναι πρώτη προτεραιότητά μας, ε, δική σας είναι εκεί η γειτονιά, χειριστείτε το εσείς το θέμα. Άρα να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε προετοιμασμένοι, να μπορούμε να έχουμε στρατηγική αυτονομία και το τι θα κάνουμε συγκεκριμένα με τις τρομοκρατικές απειλές, με την ύπαρξη τρομοκρατών στο ευρωπαϊκό έδαφος και το καθεξής. Και άλλωστε αυτό είπε και ο πρόεδρος Μακρόν το 2017, ε, κάτι που ξεκίνησε ήδη από το 2007, πολλές ευρωπαϊκές χώρες μία Βαλτική, χώρα της Βαλτικής και διάφορες σκανδιναβικές χώρες έχουν προσχωρήσει σε αυτή την προσπάθεια. Προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή ενότητα, μια κουλτούρα στρατηγική που να ε, αποτελεί αντικείμενο ευρύτερη συνένεση του τι θα πρέπει να πράξουμε στρατηγικά με αυτόνομο τρόπο, εάν τυχόν ποτέ προκύψει ανάγκη. Αυτό το και όντως με τους συναδέλφους μας από τη Ουάσιγκτον ε, ε, έχουμε την ίδια αντίληψη για την αυτονομία δράσης και αυτονομία λήψης αποφάσεων. Μπορεί να διαφωνούμε με τους Αμερικανούς για την ερμηνεία της κατάστασης, π.χ. για το Ιράν ή για το κλίμα και δεν μπορούμε να, αν έχουμε διαφορετική ερμηνεία, τότε δεν μπορούμε να έχουμε ε, πρόοδο ούτε στη λήψη απόφασης ούτε σε τίποτα. Οι Αμερικανοί δεν μας συμβουλεύονται εκ των προτέρων για κάποια απόφαση που θα πάρουν, π.χ. για την απόφαση να αποσυρθούν από τη συμφωνία. Αλλά μας συμβουλεύονται στο μετά και διαβουλεύονται μαζί μας στο μετά. Άρα έχουμε γίνει υπεύθυνοι για το Plan B, για το σχέδιο Β της Αμερικανικής κυβέρνησης και αυτό μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Αυτό Στρατηγική αυτονομία τι σημαίνει, σημαίνει να προβλέψουμε τέτοιου είδους σενάρια, σενάρια μαζί. Και αυτό θέλουμε να πράξουμε. Δηλαδή, αν είμαστε στρατηγικά αυτόνομοι, θα διαβουλεύονται μαζί μα και πριν πάρουν απόφαση, όχι μόνο μετά που την πήραν και μα φέρνουν προτετελεσμένου. Πώ δουλεύουμε με του εταίρου και του συνεργάτε μα, χωρί να ε, διακινδυνεύουμε τι αξίε μα. Στη σημερινή εποχή δεν έχουμε και επιλογή. Όταν έχουμε Ρώσους μισθοφόρους στην Αφρική, για παράδειγμα, και η Γαλλία μας ενημερώνει για τον deconflicting. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλον στην Αφρική, στη Λιβύη κτλ. Στη Συρία από το επεισόδιο του 2013 τα παραχωρήσαμε αυτά και την υπόθεση της κόκκινης γραμμής στην Τουρκία, στη Ρωσία, στο Ιράν και ούτω καθεξής σε μια περίοδο δηλαδή που εμείς οι δυτικοί, παρόλο που δεν μου αρέσει ο, ο όρος δυτικοί, αλλά για λόγους απλούστευσης, είμαστε όλο και πιο επιφυλακτικοί να χρησιμοποιήσουμε το hard power, τη σκληρή δύναμη. Τελικά η διπλωματία της κρίσης και η διαχείριση της κρίσης φεύγει όλο και περισσότερο από τα χέρια της δύση και πάει στα χέρια άλλων. Εμείς ε, έχουμε ε, όλο και λιγότερο ειδικό βάρο. Οργανώνουμε συνεχώς ε, συνέδρια, διασκέψει και γινόμαστε διαμεσολαβητές του Πούτιν, του Ερντογάν ε, για το θέμα της Λιβύης, τη Ιβυρία ή του οτιδήποτε, αλλά έχουμε χάσει και λίγο τον έλεγχο αυτή τη κατάσταση. Έχουμε μια αντιστροφή υποδείγματο. Και Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει τα πατήματά της, πρέπει να αναπτύξει μια διπλωματία διαχείρισης κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να είναι πιο γεωπολιτική. Έχουμε εκπρόσωπο εξαιρετικά δραστήριο και ενεργητικό. Αυτό είναι πολύ καλό και θα φέρει σίγουρα καρπούς να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα όθηση, τη νέα ορμή που διαφαίνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δώσουμε έμφαση σε αυτό το οποίο ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, δηλαδή οικονομική βοήθεια, διαχείριση διαπλωματικής κρίσης και διαμεσολάβηση. Μιλήσατε για το γαλλογερμανικό άξονα, ο οποίος είναι κινητήριος μοχλός για το θέμα της Ουκρανίας. Ίσως Ίσως αυτοί οι σχηματισμοί είναι coalition of the willing, είναι συμμαχίες και συνασπισμοί αυτών που βούλονται, που θέλουν, αλλά και η συμμαχία κατά του Νταές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την Ουκρανία. Όντως, εάν πρέπει αυτό το φορμάτο ad hoc να υιοθετήσουμε, γιατί όχι. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε. Αυτά λοιπόν, δεν υπάρχει και άλλη επιλογή να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους εταίρους ε, που όντω συμφωνώ δεν συμμερίζονται τις αξίες μας απαραίτητα ούτε συμμερίζονται τα δικά μας στρατηγικά ενδιαφέροντα. Ε, να μην τους αφήνουμε το πεδίο πρωτοβουλίας για να έρχονται να μας εγκαλούν μετά να διαβουλευόμαστε για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες. Είναι γεωπολιτικό το θέμα ε, που μας αφορά όλους, είτε είμαστε σύμμαχοι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία στο ΝΑΤΟ, είτε μόνο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκραντ θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, για τους ρωσικούς πυράβλους. Μεταξύ άλλων, καταδίκασε το ΝΑΤΟ την καταστρατήγηση ε, της συνθήκης ε, για τα περινικά ε, από τη Ρωσία με τις πράξεις της κτλ. Νομίζω ότι το καταδικάσαμε ομοφόνος. Τώρα, πώς θα αντιδράσουμε. Αυτό το ερώτημα τέθηκε και συνεχίζεται ο διάλογος εντός του ΝΑΤΟ. Δεν θέλουμε να βρούμε απάντηση καθρέφτη, δηλαδή να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια νέα κούρσα οπλισμών και εξοπλισμών. Όμως, θέλουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων πυλώνων της δικής μας απάντησης. Δηλαδή, από τη μία έχουμε προτάσεις ισχυρές επιστροφής σε ένα σύστημα ε, όπου η κατοχή εξοπλισμών πυρηνικών θα γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Θυμάμαι ότι στην προηγούμενη κρίση του 1969 κανείς δεν προέβλεπε τότε ότι μετά από 8 χρόνια θα είχαμε συνθήκη που θα παραγόρευε αυτή την πυραυλική ασπίδα. Άρα είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτό το μήνυμα ότι ε, πολύ γρήγορα έρχεται μια τέτοια συμφωνία. Και στο πολιτικό και διπλωματικό πεδίο Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες αλλά και στο στρατιωτικό να έχουμε αμυντικά μέσα για να σκληρύνουμε εντό εισαγωγικών το μηχανισμό μας, να τον θωρακίσουμε και να αποφύγουμε την υπερβολική ε, ε, ε, ευπάθεια του μηχανισμού μας και να έχουμε αντιπυρευλικά μέσα ή επιθετικά μέσα όχι όμως σαν να κάνουμε το ίδιο που μας έκαναν, ούτε να, να παράγουμε αυτό το οποίο κάνει η Ρωσία, αλλά για να ενισχύσουμε τη θέση μας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ε, ομιλητές για το, την εμπεριστατωμένη τους ανάλυση, για τη διαθεσιμότητά τους, για την ευγένειά τους. Να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος, που μας πλαισίωσαν καθ' τη διάρκεια του πρωινού. Ευχαριστούμε και εμείς. Και να σας υπενθυμίσω πριν ολοκληρώσουμε, 4 με 5.30 Δευτέρα, επόμενη Δευτέρα θα έχουμε την κυρία Ιζουμίνα Καμίτσου για τον αφοπλισμό αρμόδια από πλευρά ΟΗΕ. Επόμενη συνεδρίαση απόγευμα 17 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια το σύνολο όλη η μέρα της 18 Φεβρουαρίου. Τότε λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ όλους και όλες. Καλό μεσημέρι.